colleagues, good afternoon. Αγαπητοί συνάδελφοι, distinguished. καλώς ήρθατε, καλώς ορίζω και τους εκλεκτούς καλεσμένους. Πριν περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημέρας διάταξης, θα πρέπει να εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη. Σας ευχαριστώ. για τους τριλόγους και οι ανακοινώσει του Προέδρου θα γίνουν μετά την ακρόαση. Θέλω λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τους Προέδρους των τριών Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Σας έχουμε καλέσει για να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τις δραστηριότητές σας στο τελευταίο έτος. Ιδιαίτερα τον ρόλο σας σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, με τους νομοθέτες. Ε, θα θέλαμε επίσης να ξέρουμε ποιες είναι οι οργανωτικές σας προτεραιότητες για το ερχόμενο έτος και βεβαίως θα ανταλλάξουμε και απόψεις για τη μελλοντική, την επερχόμενη ε, έκθεση της ΕΣΑ την αναθεώρηση των ΕΣΑ μάλλον και διάφορες προτάσεις που θα επηρεάσουν είτε άμεσα είτε έμεσα τον ρόλο κάποιων από των υποπτικών αρχών όπως ε, το CCP και την ΕΣΜΑ. Έχουμε βεβαίω και το Brexit, έχουμε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες ε, κάποιων εποπτικών αρχών. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Επιπλέον ο κύριος Ενρία ως ε, πρόεδρος της Κοινή Επιτροπή των Τριών ΕΣΑ, έχει την κυλιόμενη προεδρία, ε, θα μας εξηγήσει πώ σκοπεύει ε, να διεκπαιρεώσει τα καθήκοντά του και ο δεύτερο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ε, του ESRB, όπω προβλέπεται το καταστατικό, υπάρχουν οι γραπτές δηλώσει για τις βασικές δραστηριότητε των αρχών που έχουν μοιραστεί, θα στα μέλη είναι διαθέσιμα υπάρχουν κάποιοι στόχοι και ε, αυτά που αναφέρει η έκθεση για τους στόχους αυτούς και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ήταν πολύ έντονη δραστηριότητα και βεβαίως ε, θα τεθεί και το θέμα των πόρων φαντάζομαι όπως πάντα εμείς σας υποστηρίζουμε οι προσδέσμες προσπάθειες δηλαδή των ESA e ε, να διεκπαιρεώσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτουμε. βεβαίω σίγουρα θα χρειαζόταν και άλλοι πόροι. Τώρα υπάρχει αυτό το νέο σύστημα που προτείνεται ε, για την αναθεώρηση της ESA. Δεν ξέρουμε αν θεωρείτε εσείς ότι αυτό, αυτή είναι η πρόταση λύνει τα προβλήματά σας, αλλά ε, σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, καλή δουλειά όμως, ε, στα πλαίσια, σε ένα πνεύμα αγαστής συνεργασίας. Βεβαίως δεν συμφωνούμε πάντα για όλα τα ζητήματα, αλλά έως τώρα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, Τώρα έχουμε τα πρώτα σχόλια. Θα δώσω το λόγο στον ε, Ανδρέα Ενδρία που έχει 12 λεπτά στη διάθεσή του για να μιλήσει και ως πρόεδρος της, ε, Επιτροπ... της Κοινής Επιτροπής και ως αντιπρόεδρος της ESRB. Ή Ανδρέα, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, ο Ανδρέα λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ την τελευταία έκθεση για τον διατομιακό κίνδυνο έχουμε υπογραμμίσει τρία σημεία ανησυχίας. UK's withdrawal e ε, παρουσίας κινδύνων και χαμηλή ε, παραγωγικότητα και κερδοφορία. Υπάρχουν και αρκετά θέματα τα οποία τίθενται σε επίπεδο εποπτείας λόγω του Brexit και αυξάνουμε τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για τους πιθανούς κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Είμαστε προσεκτικοί επίσης και για την κατάσταση σε πιστοτικά ιδρύματα και σε ποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει γενικότερα τις αγορές και να προκαλέσει ζημίες για τους επενδυτές. Υπάρχει επίσης και θέματα, υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ε, ασφάλειες. κάναμε μια ημερίδα καταναλωτών όπως την ονομάσαμε στην Πράγας και εκεί υπήρξαν ε, πολλοί χρήστες ε, των υπηρεσιών που παρέχουν τα πιστοτικά και ασφαλιστικά ιδρύματα και προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε με καλύτερο τρόπο τους άμεσα εμπλεκομένους. Ε, υπήρξαν αρκετές ιδέες και νομίζω ότι περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και συνεισφορές και από δική σας πλευράς. Επίσης ε, έχουμε προχωρήσει στη συλλογή, στην παροχή τεχνικών συμβουλών για τα PRIBS. Υπάρχουν ε, θέματα που τίθενται και από τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως οι συζητήσεις ε, για τον αυτοματισμό στις χρηματοπιστωτικές συμβουλές, όπως επίσης και τη διαχείριση των λεγόμενων big data. Υπάρχουν κίνδυνοι βέβαια ακόμα για τους καταναλωτές. Από τη μία η προσωποποίηση, η εξατομίκευση των συμβουλών περιορίζει τις δυνατότητες συγκρισιμότητας ε, τις οποίες θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής. Ταυτόχρονα αυτού του είδους οι καινοτομίες ε, μπορεί να ε, δημιουργήσουν δυνατότητες νέων κερδών από πλευρά των αλλά από την άλλη οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πλήρη κατανόηση των πληροφοριακών δελτίων. Θα πρέπει λοιπόν, εφόσον εντοπίσαμε τους κινδύνους, να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των μέτρων τα οποία έχουμε αποφασίσει ήδη για την μετρίασή τους πέρα από την ολοκλήρωση της εντολής μας της αρχικής υπάρχουν αρκετές ε, εξωτερικές περιπτώσεις όπως τα Panama Papers και άλλες περιπτώσεις οι οποίες δημιουργούν ανάγκες για μεγαλύτερη ανάλυση ε, και καλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης και αξιολόγησης κινδύνων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να ανταλαμβάνουν όλα αυτά υπόψη όταν ε, λαμβάνουν υπόψη επίσης και το θέμα της, ε, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος έτσι ώστε η λεγόμενη κίνδυνη MLTF είναι σε αποδεκτό μέχρι στιγμής επίπεδο. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος ε, βασίζεται στα ευρήματα στα πλαίσια της έρευνας για τα Panama Papers, είναι η βελτίωση της ανταλλαγής ενημέρωσης και στοιχείων ανάμεσα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μεγαλύτερη ασφάλεια και βεβαιότητα και στον τομέα αυτό μέσω ισχυρότερης συνεργασίας. Επαναλαμβάνουμε επίσης ε, την ανησυχία μας ε, και για ε, την εφαρμογή του iFrest 9 για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε ευρύτερους διεθνείς ομίλους. Θέλουμε να υπάρξει σωστή διαιτησία σε σχέση με την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών, γιατί έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα έχουμε χαμηλότερα από τα επιθυμητά επίπεδα προστασίας των επενδυτών. Στα πλαίσια τώρα της προστασίας των καταθετών καταναλωτών, οι ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν είναι, θα έλεγα, δύσκολες στη χρήση τους. Υπάρχει ανάγκη, εν πάση περιπτώσει, για βελτίωση της στρατηγικής επεξεργασίας των σημείων τα οποία συλλέγουμε στα πλαίσια της παρούσας κατάστασης. Σχετικά τώρα με τα τραπεζικά θέματα έχει υπάρξει βελτίωση σε σχέση με τους ισολογισμούς των τραπεζών. Ε, τα, ε, τα επίπεδα κεφαλαίων έχουν επίσης βελτιωθεί, όπως επίσης έχει βελτιωθεί και το χαρτοφυλάκιο των πιστοτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ε, ποιοτικό. Μιλάμε για 9 δις περίπου ευρώ και Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες βέβαια. Εκεί όπου υπάρχει υψηλή ρευστότητα αγορός, ε, ε, ε, ρευστότητα προσφοράς, τα επίπεδα απόδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των δευτερευουσών αγορών και σε σχέση με τη διαχείριση των MPLs σύμφωνα και με τις εθνικές ρυθμίσεις. Το IRFS 9 από την αρχή του 2018 θα προκαλέσει αρκετές αλλαγές και περιμένουμε τις νέες εκθέσεις για την αξιολόγηση του νέου πλαισίου έτσι ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σωστά προετοιμασμένες. Τώρα για την δυνατότητα απορρόφησης απολειών, ζημιών. οι ευρωπαϊκές συστημικού ενδιαφέροντος τράπεζες ήδη είναι στο επίπεδο ή είναι πολύ κοντά στο να είναι στο επίπεδο ε, των νέων ε, παγκόσμιων ρυθμίσεων που θα τεθούν σε ισχύ από το 2019. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Για να υποστηρίξουμε τις απαιτούμενες αλλαγές ε, στα πλαίσια της δυνατότητας απορρόφησης ζημιών, θα πρέπει να τελειώσει η διαδικασία αλλαγών στα EBRD και να επιτευχθούν οι στόχοι MREL. Έτσι θα βελτιωθεί το κλίμα της αγοράς και έτσι θα ρυθμιστεί και το θέμα των ζημιών που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να απορροφηθούν απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα σαν επενδυτές να αξιολογήσουμε σωστά τις, ε, τα αρνητικά των τραπεζών. Η Εποπτική Αρχή επίσης δημοσίευσε και μία έκθεση για τις επιπτώσεις των προτινόμενων αλλαγών όπως του ποσοστού της μόχλευσης και τον MREL. Προσπαθήσαμε να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για την δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι εργασίες της Επιτροπής της Βασιλείας βρίσκονται πάρα πολύ κοντά σε επίπεδο ολοκλήρωσης. Τα διεθνή στάνταρ, δηλαδή θα καθοριστούν πλήρως και αυτό θα μας ε, χρησιμεύσει σαν πλατφόρμα και για την διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αντίστοιχων ρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σε συνεργασία με την ΕΣΜΑ έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού πακέτου λόγω των ε, επιμέρους διαφορών που ισχύουν στις διάφορες χώρες Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα κοινό πλαίσιο με κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στα επιχειρηματικά πρότυπα. Η αύξηση της αναλογικότητας σε επίπεδο κατευθυντήριων αρχών και συμμόρφωσης είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε υπόψη για το PSD2 ήταν προτεραιότητα της προσπάθειάς μας, οι προτάσεις για τα RTS, για την ασφαλή επικοινωνία ήταν ε, κάτι από τα πιο δύσκολα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί. Λάβαμε πολύ διαφοροποιούμενα σχόλια από τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους και έπρεπε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στον ανταγωνισμό από τη μία και την ασφάλεια και βεβαιότητα από την άλλη. Και γι' αυτό ζητάμε να τροποποιηθεί η RTS σε συγκεκριμένους τομείς. Τώρα για τη διατήρηση των παραδοσιακών πιστοτικών δραστηριοτήτων δημοσιεύσαμε εμείς ε, μία έκθεση για τα FinTech και τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις τραπεζικές δραστηριότητες. Επίσης τα καθεστωτα SM S-Boxing και γενικότερα θέματα προστασίας των καταναλωτών όπως επίσης και την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών και των μέσων IT έτσι ώστε να προστατεύονται από εξωτερικές επιθέσεις εις βάρος των τραπεζών και των καταναλωτών. Επίσης και στον τομέα της τυπλοποίησης είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει και τις συστάσεις για την ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου πακέτου απαιτήσεων κάτι το οποίο θα καταστήσει ε, ξεκάθαρα το ποιες επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες τύπου MIFED. Θα πρέπει επίσης ε, να ελεγχθεί και το θέμα του κοινού δικτύου και του κοινού επίπεδου ελέγχου στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις εσωτερικών μοντέλων, ενέργειες back-to-back, back to back όπως επίσης και ε, διαδικασίες σχετικά με τις εκαθαρίσεις τραπεζών και εγγυήσεις καταθέσεων. Υπάρχει και το θέμα της μετακόμισης της EBA, της, ε, της εποπτικής μας αρχής. Είναι κάτι το οποίο μας ε, δημιουργεί προβλήματα, δημιουργεί αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες Ήδη από την αρχή του καλοκαιριού έχουν υπάρξει πάρα πολλές παρετήσεις λόγω της προφανούς μετακίνησης. Είναι κάτι το οποίο θα απαιτήσει πάρα πολύ χρόνο και θέλουμε χρόνο για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις συνέπειες αυτής της μετακίνησης. Ταυτόχρονα η τροποποίηση και του τρόπου λειτουργίας μας έτσι ώστε να αρμόζει περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το απαιτεί περαιτέρω χρονικό διάστημα. Thank you very... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Ανδρέα. Τώρα περνάμε στον κύριο Μπερναρντίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σήμερα θα εστιάσω στο πώς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την προστασία των κανοντών, να υπάρξει μια θυμιστική σύγκληση και να έχουμε μια χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Στο τέλος αναφερθώ στις μελλοντικές ε, τάσεις και ευκαιρίες. Παρά την, το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον όπου έχουμε ιστορικά χαμηλά επιτόκια, η εφαρμογή της οδηγίας περιφερειακότητας υπαρχών 2 έγινε επιτυχώς ε, κυρίως λόγω, στο, κυρίως λόγω των μεταβατικών περιόδων και της αναλογικότητας. Σήμερα μπορώ να πω ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος των ασφαλιών ωφελείται από αυτό το εύρωστο καθεστώς και είναι πολύ ισχυρότερος. Η πιο συντονισμένη εποπτεία είναι αναγκαία για να μην υπάρχει ρυθμιστικό αρμπιτράζ. Το τελευταίο έτος αναπτύξαμε περαιτέρω το βιβλίο των ορθών πρακτικών μας με βάση την οδηγία για την φερεγγιότητα και βεβαίως συνεχίσαμε τις επαφές με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Ε, έτσι, ανοιχνεύσαμε διάφορα ζητήματα που αφορούν τα επιχειρηματικά μοντέλα που εκμεταλλεύονται το καθεστώ ελευθερίας παροχής υπηρεσιών που σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησε σε χρεοκοπία ασφαλιστικών εταιριών ε, κατά το οποίο ζημίωσε τους συμβαλόμενους. Γι' αυτό ενισχύουμε την ρυθμιστική συνεργασία σε διασυνοριακές ε, επιχειρήσεις, ε, δημιουργώντας ακριβώς ε, τις διασυνοριακές αυτές πλατφόρμες που συντονίζει η αρχή μας. Πολλές τέτοιες έχουν δημιουργηθεί και είναι επιτυχής και έτσι παρεμβαίνουμε πολύ νωρίτερα και περιορίζουμε τις περαιτέρω καταστροφικές συνέπειες στους Ευρωπαίους ασφαλισμένους. Οι δραστηριότητες μας σε Ρουμανία και Βουλγαρία για τον έλεγχο των ισολογισμών δείχνουν πως η ανάληξη κινδύνων από τις ε, ασφαλιστικές εταιρείε θα πρέπει να επιτηρείται καλύτερα και να τηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έγιναν επίσης επισκέψεις αρμόδιες αρχές και τεχνικές αναλύσεις και έτσι είδαμε πώς υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές στις διάφορες χώρες ανάλογα με τα εσωτερικά μοντέλα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείε να λάβουν αυθαίρετες αποφάσεις όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο κάλυψης των μοντέλων τους. Και εδώ πέρα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να διασφαλίσουμε μια αριθμιστική σύγκληση όσον αφορά την προστασία των ε, καταναλωτών. Καλωσορίζουμε την απόφαση της ε, Κομισιόν ε, να λάβει υπόψη στην σχετική οδηγία τις περισσότερες ε, συστάσεις μας. Όμως απογοητευτήκαμε επειδή βλέπουμε πως οι πληρωμές ε, τρίτων μερών δεν έχουν περιληφθεί στον κατάλογο των χαρακτηριστικών περιπτώσεων αντικρώμενων συμφερόντων. Η ε, θεματική παρακολούθησή μας όσον αφορά τις αμοιβές στις ασφαλιστικές εταιρείε ήταν η πρώτη πανευρωπαϊκή τέτοια ανάλυση για ζητήματα προστασίας των καταναλωτών. Για να ενισχύσουμε επιπλέον ε, την εικόνα μας για την ε, αγορά των συντάξεων σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρόσφατα ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση για τις απαιτήσει ε, στατιστικών αναφορών για τα συνταξιωτικά ταμεία. Όσον αφορά λοιπόν τις ατομικές συντάξεις, καλωσορίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να εισαχθεί το πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικής σύνταξης, το οποίο έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει μια ενιαία τέτοια αγορά προς όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Θεωρούμε πως ο ρόλος μας θα είναι ουσιαστικός για να διασφαλιστεί η χρήση ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας και να υπάρξει αποτελεσματική εποπτεία. Η Ευρώπη θα πρέπει να αφιερώσει τους απαραίτητους πόρους σε αυτό. Τον Δεκέμβριο του 2016 δημοσιεύσαμε τα αποτελέσματα των τελευταίων stress test των ασφαλιστικών εταιριών και κάναμε μια εκτίμηση των αδυναμιών του κλάδου των ε, ασφαλιών στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων. Είχαμε κάποιες συστάσεις και παρακολουθούμε την εφαρμογή τους. Έχουμε τώρα το δεύτερο στρες τεστ το οποίο λαμβάνει η χώρα και θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα στο τέλος του έτους τον Ιούλιο. Επίσης εκδώσαμε μια γνωμοδότηση η οποία απευθύνεται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για το ελάχιστο ανάκτηση ανάκτησης ε, και λύσης των εταιριών, ειδικά σε περιπτώσεις διασυνοριακών επιχειρήσεων. Θα πρέπει έτσι να αποφεύγεται το κόστος εκείνο το οποίο δεν είναι απαραίτητο, το οποίο προκύπτει από διαδικασίες αποφάσεων, ε, λήψης αποφάσεων οι οποίες δεν είναι συντονισμένες. Επιπλέον, δεδομένων των ουσιαστικών διαφορών σε χρηματοδότηση, πεδίο εφαρμογής και κάλυψη, η ΕΟΠΑ θα εξετάσει την δυνατότητα ενός ελάχιστον αρμονισμένου πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το μέλλον. Ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα απαιτεί το να παραμείνουμε σε εγρήγορση. Παραδείγματο χάρη όσον αφορά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποσυρθεί, η ΕΟΠΑ δημοσίευσε μια γνωμοδότηση για να στηρίξει τις εθνικές εποπτικές αρχές όσον αφορά την μετακόμιση επιχειρήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, θα πρέπει να μην αποδεχόμαστε εταιρείε γραμματοκιβώτια. Στο μέλλον απαιτούνται τολμηρότερα βήματα για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και την ολοκλήρωση της αγοράς των χρηματαγορών. Στο πλαίσιο αυτό, καλωσορίζουμε την πρόταση Κομισιόν για την αναθεώρηση της εποπτικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης. Σκοπεύουμε λοιπόν να αναπτύξουμε στρατηγικά εποπτικά σχέδια και να ενδυναμώσουμε τις ανεξάρτητες αξιολογήσει των ιστορικών μοντέλων. Επιπλέον, καλωσορίσαμε την πρόταση για να περιληφθεί η βιωσιμότητα αλλά και η τεχνολογική και στην εντολή μας. Οι εποπτικές αρχές έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν ε, έτσι ώστε οι καταναλωτές θα μπορούν να ωφελούνται από την καινοτομία, παραμένοντα προστατευμένοι. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά τι εσυνοριακέ δραστηριότητε, απαιτείται μια ακόμη πιο στιβαρή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η δυνατότητα οι υπηρεσίε να αποκτούν διαβατήριο σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υποπτία του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα πρέπει η ΕΟΠΑ να έχει την εντολή να παρεμβαίνει πιο δυναμικά για να γίνει αυτό, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να ειδοποιούν την ΕΙΟΠΑ εγκαίρως στην περίπτωση στην οποία οι εταιρείε ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες που μπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις επιπλέον σε σχέση ε, με την ε, εποπτική ανεξαρτησία και τα δικό συμφέροντα θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος μας. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ε, δημιουργία των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ε, για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον προστασία του καταναλωτή και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και είμαι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για την αναθεώρηση του κανονισμού μα για να έχουμε ανεξαρτησία και λόγοδοσία και μια ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλιστικών εταιριών και των συντάξεων με αυτά ωφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, ο κύριος Μαϊζόρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Ρομπέρτο, αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω εν συντομία για τις δραστηριότητε της ΕΣΜΑ του τελευταίους 12 μήνες και τις μελλοντικέ προκλήσεις για την κεφαλαία αγορά, την ευρωπαϊκή και την ΕΣΜΑ. Θα ήθελα να αναφερθώ να ευχαριστήσω καταρχήν τα, τα μέλη τη Επιτροπή για, για το συνεχή και επικοδομητικό διάλογο που έχουμε την ΕΣΜΑ. Είμαι πεπισμένο ότι η συμμετοχή τη ΕΣΜΑ ε, έχει συνεισφέρει στην πολιτική συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σε αυτό το κοινοβούλιο. Θα αναφερθώ στου τέσσερι βασικού τομεί δραστηριότητα τη ΕΣΜΑ. Ε, ο νέο του, ο κανόνας ανάλυση κινδύνου άμεση εποπτεία μεταξύ άλλων. Γι' αυτό το σκοπό θα επικεντρωθώ σε δύο σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ευρωπαϊκούς τίτλους. Καταρχήν η εφαρμογή και δεύτερο το Brexit. Ε, Πρώτα η εφαρμογή, η εφαρμογή του MIFID 2 βεβαίως. Ε, θέλω να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό αλλά και ταυτόχρονα ε, δύσκολο και απαιτητικό σε πέδο πόρων είναι το έργο αυτό της εφαρμογής της MIFID. Η εφαρμογή του MIFID 2 θα απασχολήσει τη ρυθμιστική, τις ρυθμιστικές αρχές για πολύ καιρό. Έχουν γίνει μεγάλες οπάδες από την ΕΣΜΑ έτσι ώστε να φτάσουμε σε εφαρμοστικά μέτρα έγκαιρα. Τα πιο πρόσφατα αφορούν ε, τις υποχρεώσεις ε, σε ό,τι αφορά τα παράγωγα που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικούς μήνες. Η εφαρμογή του MIFID 2 δείχνει ότι ο το εγχειρίδιο με τους ενιαίους κανόνες πρέπει να συμπληρωθεί. Τους τελευταίους 12 μήνες λοιπόν η ΕΣΜΑ έχει προετοιμάσει μια από γραμμές ε, και Q&As για να απαντήσει σε ερωτήματα από τις αρμόδιες αρχές και, και παράγοντες της αγοράς ώστε να υπάρξει μια συνεχή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που τίθεται σε ισχύ. Ένα μέρο αυτή τη δουλειά σύγκληση σχετίζεται με τι προσπάθειε τη ΕΣΜΑ να ενισχύσει την προστασία του καταναλωτή, κάτι που είναι από του βασικού σκοπού τη ολόκληρη μεταρρύθμιση MIFID. Επιπλέον, εγώ είμαι αισιόδοξο για το κατά πόσο μπορούμε να ε, ε, επιχειρήσουμε στο νέο πλαίσιο σε λιγότερο από τρει μήνε από σήμερα. Βεβαίω δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το μέγεθο και την περιπλοκότητα αυτού του σχεδίου και βεβαίω μπορεί να προκύψουν προβλήματα στην αρχική επιχειρησιακή περίοδο. Η ΕΣΠΑ αναγνωρίζει ότι είναι πολλέ οι προκλήσει για όλου του εμπλεκόμενου και όλα αυτά τα ζητήματα θα τα εξετάσουμε με, τους, ε, με τα υπάρχοντα εργαλεία καθώ θα προχωράει η εφαρμογή. Από εκεί και πέρα θέλω επίση να την προσοχή σα ε, στου περιορισμού σε επίπεδο πόρων ε, σε επίπεδο ΕΣΜΑ. Αυτό αναφέρθηκε ήδη από τον Ρομπέτο. Χρειάζεται λοιπόν προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τα σχέδια. Χρειάζονται προτεραιότητε. Είχαμε μια πρόσφατη συμφωνία με τα NCAs έτσι ώστε ε, τα ζητήματα διαφάνειας να ε, εφαρμοστούν προοδευτικά από τον Ιανουάριο του 2018. Τώρα θα αναφερθώ στα ζητήματα που αφορούν το Brexit. Αυτά σχετίζονται με όλες τις βασικές δραστηριότητες της ΕΣΜΑ. Καταρχήν να σας πω ότι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά συμμετέχονται στην αγορά που πρέπει να μετακατασταθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ευρώπη των 27 για να να έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά δημιουργεί ανησυχίες σε ό,τι αφορά τις διατησίες, τις ρυθμιστικές μεταξύ των, χωρών, των 27 χωρών ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν αυτές τις επιχειρήσεις. Χρειάστηκε, λοιπόν μια έγκαιρη απάντηση. Εμείς προτιμάσαμε μια γνωμοδότηση γενική και τρει επιμέρου γνωμοδοτήσει. Ασχολούμαστε με τη σημεία κλειδιά που έχουν να κάνουν με το outsourcing και την ε, εξουσιοδότηση στι τρίτε χώρε. Βασιζόμαστε κυρίω στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, την υπάρχουσα. Δίνουμε κατάσταση και τι γραμμέ προ τι NCAs που αυτή τη στιγμή λαμβάνουν πολλά αιτήματα από διάφορε οντότητε που θέλουν να μετεγκατασταθούν. Από εκεί και πέρα το ε, Brexit μπορεί να δημιουργήσει και σημαντικού κανόνε σε πέδο ε, σταθερότητα. Ιδιαίτερα εφόσον δεν υπάρχει κάποιο διακανονισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ΕΣΜΑ παρακολουθεί στενά τα ζητήματα όπου θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερου κινδύνου για του επενδυτέ και για τι αγορέ στο σύνολό του. Μαζί με τι άλλε αρμόδιε αρχέ συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να μετριάσουμε αυτού του κινδύνου. Επίση, το Brexit έχει δημιουργήσει και ευρύτερε πολιτικέ συζητήσει και αυτή την Επιτροπή για το κατά πόσο το υπάρχον μοντέλο ισοτιμίας με τις τρίτες χώρες είναι, είναι κατάλληλο. Εμείς έχουμε αρχίσει να εξετάσουμε τις κατέρες γραμμές ε, για την έγκριση των ε, ε, πιστο, πιστοληπτικών ε, αρχών τρίτων, αρχών, αρχών μάλλον αξιολόγησης. Βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει σε επίπεδο Επιτροπή σε ό,τι αφορά τον κανονισμό ΕΜΙΡ και χαίρομαι που έχουν, που έχει υποληθεί πρόταση κάποιες ε, ρυθμιστικές εξουσίες, εποπτικές εξουσίες για τις τρίτες χώρες και τα CCPs ε, δίνονται πλέον στην ΕΣΜΑ. Θα πρέπει βεβαίως η ΕΣΜΑ όχι μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις ό,τι αφορά τις ισοδυναμίες, αλλά και τα benchmarks των τρίτων χωρών ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να έχει η ΕΣΜΑ εξουσία και για κάποιους, ε, κάποιες χρηματαγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ πραγματικά θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να το συζητήσω αυτό μαζί σας, καθώς και άλλα στοιχεία της πρόσφατης ανθεώρησης της ΕΣΜΑ εντός των επόμενων εβδομάδων και μηνών. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις, στην εξέλιξη της ε, Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς, της Κεφαλαϊκής Ένωσης. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά ε, την, τις ε, υπηρεσίες ε, τις επενδυτικές θα λάβει χώρα και ένα έργο αξιολόγησης ομοτήμων θα συνεχίσουμε το έργο αυτό, διότι μας οδηγεί σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για κάποια κράτη-μέλη και την ασυνέπεια σε ό,τι αφορά τις πρακτικές εποπτείας. Αυτά και άλλα εργαλεία εποπτικής σύγκλησης που θα βελτιωθούν με την αναθεώρηση της ΕΣ θα βοηθήσουν στην ΕΣΜΑ έτσι ώστε να βελτιωθεί η προστασία του καλωτήκα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι αφορά την κεφάλαια αγορά, η ελευθερία του να εγκατασταθεί κάποιο σε, μια χώρα και να υπάρχει υπηρεσία σε όλε δίνει πολλέ πολλές δυνατότητε. Αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε. Ένα στοιχείο τη CMU πρέπει να αναφέρουμε εδώ και που συνδέεται με την εποχή μετά τη κρίση, όταν δημιουργήθηκε η ΕΣΜΑ, είναι οι αναφορέ και η συλλογή δεδομένων. Η ΕΣΠΑ έχει αφιερώσει πολλού πόρου για να δημιουργηθούν πολλά συστήματα αναφορών. Ταυτόχρονα θέλουμε να αποφύγουμε τι επικαλύψει και να βασιστούμε στι υπάρχουσε απαιτήσει. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τα γενναία βήματα έτσι ώστε να διατηρήσουμε το momentum που υπάρχει ε, με βάση τι πρωτοβουλίε που έχουν ήδη ξεκινήσει. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να ενισχύσουμε τι ευρω... ευρω... ευρωπαϊκέ κεφαλαίε Πρέπει να σα σας πω ότι η ΕΣΜΑ θα υποστηρίξει αυτού του στόχου και αναμένω μια στενή συνεργασία για αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και του ε, τρει προέδρου και τώρα θα ξεκινήσει ο διάλογος. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Μπούρχετ Βάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας εδώ και καιρό ζητούσε μια αλλαγή του κανονισμού της ΕΖΑ. Τώρα έχουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε εμπειρία πλέον 6,5 ετών. Εσείς ε, στις υπηρεσίες σας και εμείς από την συνεργασία μαζί σας και οπωσδήποτε έχει φτάσει η στιγμή για μια μετεξέλιξη του status quo βεβαίως. Εμείς ως νομοθέτες πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και πιθανώς ε, διεύρυνση των εντολών σας και να υπάρξει ε, μια καλύτερη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των διαχωριστικών γραμμών των διαφόρων εποπτικών αρχών. Και έχω άρα μια ερώτηση προς τον κύριο Ανδρέα Ενρία πρώτα και μετά προς τον κύριο Μαγιόρ. Η ε, ερωτήση μου είναι εξής. Φαίνεται πως ο Στίβεν Μαγιόρ αυτή τη στιγμή ίσως είναι ευτυχέστερος από εσάς τους ε, τρεις καθώς έχει άμεση εποπτική αρμοδιότητα και περισσότερα δικαιώματα και θα έχει περισσότερα δικαιώματα άμεσης παρέμβασης. Ε, βεβαίως, όπως γνωρίζετε, εμείς θέλουμε να υπάρχει ένας ε, κανονισμός ανακλάδο για τον τομέα, δηλαδή των τραπεζών της ασφάλισης και των αγορών, γιατί ο κάθε κλάδος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και απαιτεί τομεακή και περιφερειακή ε, εμπειρία. Εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή με την πρόταση της Κομισιόν να μην γίνει κάτι τέτοιο με την ΕΣΜΑ. Και μετά μία ερώτηση για τους άλλους δύο κυρίους. Ξέρετε ότι συνεχώς με απασχολεί το θέμα της αναλογικότητας. Η πρόταση της ε, Κομισιόν εδώ πέρα κάπως υστερεί και θα έπρεπε να έχει μια καλύτερη αιτιολόγηση και ίσως να υπάρξει περισσότερη διαβούλευση. Πώς μπορούν να γίνουν περισσότερα για να υπάρξει περισσότερη αναλογικότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάλτς. όσον αφορά τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Οπωσδήποτε είμαστε σε άλλον πλανήτη γιατί έχουμε ήδη την Τραπεζική Ένωση που έχει ήδη συγκεντρώσει τα εποπτικά καθήκοντα. Οπότε λογικό είναι να απαιτείται ανάλογο συγκεντρωτισμός και στην κεφαλαία αγορά. Οπότε δεν βλέπω κάποια σύγκρουση μεταξύ των δύο. Ε, βλέπω θετικά κάποιες προτάσεις. Ξέρετε, το συζητάμε εδώ και καιρό. Έχουν υπάρξει κάποια αποπτικά καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στην τραπεζική αρχή που είναι κάπως δύσκολο να εξασκηθούν π.χ. αυτά τα οποία αφορούν τα stress ή την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου ή περιπτώσεις διαμεσολάβησης. Και η πρόταση της Κομισιόν νομίζω δημιουργεί διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να ασκήσουμε αυτά τα καθήκοντα. Και για να είμαι ειλικρινής, η διοίκησή μας έχει στηθεί γύρω από την έννοια της πίεσης ε, θα έλεγα, κάτι το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε. Οπότε μια διαφορετική προσέγγιση νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Για την αναλογικότητα γνωρίζω ότι ναι, Πράγματι γίνονται κάποιες σκέψεις, ε, είπα και πριν ότι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στους δικούς μας κλάδους, π.χ. στον τομέα των αναφορών, του πυλώνα 2 ή και πυλώνα 3 βεβαίως. Ε, περισσότερες τράπεζες ε, παραπονιούνται για τον αριθμό των δηλώσεων που πρέπει να κάνουν. Εμείς προτείνουμε να μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για να μειωθεί το ρυθμιστικό βάρος χωρίς να διαφοροποιούνται οι απαιτήσει ε, ανάλογα με το μέγεθος και την περιπλοκότητα. Σας ευχαριστώ κύριε Μπάλτς. Ε, θα προσπαθήσω να καλύψω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα για την πρόταση της ε, Κομισιόν. Το πρώτο το οποίο είναι θετικό νομίζω είναι ότι υπάρχει αυτή η ολιστική προσέγγιση η οποία εξετάζει και την προληπτική πτυχή και την εποπτεία Νομίζω ότι αυτό ήταν θετικό. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες ε, και πάλι όπως είπε ο Ανδρέα, στις ασφάλειες ε, δεν έχουμε μια ασφαλιστική ένωση, οπότε οπωσδήποτε καλώς ορίζουμε το ότι υπάρχουν προτάσεις ε, να δοθεί μια ισχυρότερη εντολή στην ΕΙΟΠΑ για να υπάρξει μια σύγκληση. Εμείς οπωσδήποτε μπαίνουμε σε αυτόν τον τομέα της εποπτείας και όσο περισσότερα βλέπουμε νομίζω λέμε ότι μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Για να είμαι ειλικρινής, απαιτείται περισσότερη ουσία, μια ισχυρότερη εντολή δηλαδή. Και όπως είπα, ειδικά σε περιπτώσεις ε, διασυνοριακών επιχειρήσεων όπου έχουν διαφορετικά συμφέροντα η χώρα προέλευση και προορισμού και η μόνη φωνή που περασπίζεται τους ε, Ευρωπαίους ασφαλισμένους είναι η ΕΟΠΑ. Τρίτον για την αναλογικότητα Γνωρίζετε ότι βεβαίω αυτό είναι μια μάχη που δίνει από την αρχή της ε, φερεγγιότητας 2. Έχουμε προχωρήσει πολύ στη ρυθμιστική πλευρά. Ε, π.χ. στις ε, αναφορές έχουμε προχωρήσει πολύ. υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο συχνά υποτιμάμε. Η εποπτεία. Μεγάλο κομμάτι δηλαδή της αναλογικότητας πρέπει να υπάρξει και στο πώς εφαρμόζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις ε, αναλογικότητας ναι, στο εποπτικό σκέλος. Π.χ. τώρα αυτή τη στιγμή εξετάζουμε συγκριτικά τις ε, κύριες λειτουργίες του συστήματος ε, διακυβέρνησης και βλέπουμε ότι οι εθνικές αρχές ακολουθούν πολλές και διαφορετικές πρακτικές για την αναλογικότητα. Αυτό λοιπόν αφορά όχι μόνο τον κανονισμό, αλλά την ε, τη ρύθμιση, αλλά την εφαρμογή και εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ομοιομορφία. Ναι, συντομία, ο κύριος Μπάρτ θέλει να μιλήσω και για την αναλογικότητα φαντάζομαι. Θα είμαι σύντομος. Ε, ακούστε, αυτό που έχει σημασία εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από την εφαρμογή για να βελτιώσουμε περαιτέρω την υπάρχουσα νομοθεσία. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευτυχή με τις βελτιώσεις στο ΕΜΙΡ, το ΕΜΙΡ 2.0. Ε, εξετάζουμε εδώ τα στοιχεία. Ποια είναι η επιβάρυνση για τις πιο μικρές οντότητες. Μπορούμε να τις ε, εξαιρέσουμε. Μήπως αυτό θα δημιουργήσει όμως ε, ε, προβλήματα, διότι υπάρχει ένα θέμα λογικότητας. Ε, έχει νόημα με βάση τον πιο μικρό ποσοστό κινδύνου που παρουσιάζουν οι μικρότερε οντότητε. Πρέπει πάντω να αξιολογούμε τακτικά την νομοθεσία μα και με βάση εμπεριστατωμένα στοιχεία να αλλάζουμε τα πράγματα και να βελτιώνουμε βεβαίω την νομοθεσία. το, το άλλο θέμα είναι τα δεδομένα. Βεβαίω, πολύ περίπλοκο το θέμα των δεδομένων. Ε, για τι μικρέ οντότητε και αυτό είναι πολύ επιβαρυντικό ε, και οποιαδήποτε ευθυγράμμιση θα βοηθούσε εδώ. Ε, ναι, Περβόν Μπερέζ, ευχαριστώ. Είστε εδώ για να παρουσιάσετε το πρόγραμμα εργασιών σα. Θα υπάρξουν πολλά ερωτήματα, φαντάζομαι, για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά. Ε, σε αυτό το πνεύμα θέλω να επανέλθω στο θέμα τη διακυβέρνηση, διότι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Με βάση τη δική σα εμπειρία, του καθενό από εσά, με βάση τι ε, ε, εξουσίες που έχετε, τις αρμοδιότητές σας, σε αυτή τη δομή των διαφόρων οργανισμών, τι είναι αυτό που σας λείπει περισσότερο σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, σε επίπεδο εξουσιών. Πιστεύω ότι η πρόταση τη Κομισιόν πρέπει να σε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα και σε επίπεδο διαμεσολάβηση και κάτι άλλο. Είστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι δίνετε μια κάποια σημασία στον διάλογο που έχουμε μαζί σας και με βάση τα αποτελέσματα ε, και τη εμπειρία που έχουμε αποκομίσει σε αυτό το διάλογο, το Κοινοβούλιο έχει παίξει και ρόλο στον ορισμό, ε, ορισμό στι θέσει αυτέ. Αν θεωρείτε ότι η πρόταση τη Κομισιόν είναι ικανοποιητική, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική, αλλά πείτε μα κι εσεί. Γκάμπριελ, ευχαριστώ πολύ κυρία Μπερέζ. Δύο-τρία πράγματα να πω για τη διακυβέρνηση. Εάν δείτε τα ρυθμιστικά ζητήματα και το πώς ε, προχωράμε ε, στις τρεις αυτές ε, στους τρεις αυτούς οργανισμούς, με διαφανή τρόπο πιστεύω, έχει λειτουργήσει αρκετά καλά το σύστημα. Εκεί όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούμε είναι στο επίπεδο της εποπτείας. Και όσο αυξάνεται η εντολή μα σε αισθήματα εποπτεία, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογέ σε επίπεδο διακυβέρνηση. Διότι δεν μπορούμε να πάρουμε τι αποφάσει που, που χρειάζονται έγκαιρα ε, σε αυτήν την παρούσα διαδικασία που προβλέπετε. Και για το τρίπ δεν μπορούσατε να πάρετε αποφάσει, λέει η κυρία Μπέρε. Ναι, έχετε δίκιο. Υπήρξε απόκληση απόψεων από το ένα οργανισμό στον άλλον. Αλλά αυτό ήταν όμως ε, ε, εξαιρετική περίπτωση. Ε, πρέπει να γίνουν προσαρμογές λοιπόν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα εποπτείας. Τώρα για τη διαμεσολάβηση. Ε, θα αναφερθώ και στην παραβίαση του κοινωτικού δικαίου. Έχουμε εμπειρία από καταστάσεις διαμεσολάβησης. Τώρα για την παραβίαση, ακούστε, αυτό είναι ατομική βόμβα, έτσι ας είμαστε ειλικρινείς, ε, δεν μπορεί να προκύψει αυτό το πράγμα, δηλαδή η παραβίαση της κοινωνικής νομοθεσίας από τις οπτικές αρχές. Χρειαζόμαστε πιο πολλά στοιχεία για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πιο ισχυρές αποφάσεις από ευρωπαϊκής πλευράς. Δηλαδή δεν μπορεί το θέμα της των, ε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας να θεωρηθεί η πανάκια λύσει τα προβλήματά μας. Να δώσω κάποια παραδείγματα για τη διαμεσολάβηση. Αναφερθήκατε στη διαμεσολάβηση, κυρία Μπερέ, και πολύ σωστά, διότι είναι ένα σημείο κλειδί. Ε, είχαμε μια σειρά από περιπτώσει όπου γνωρίζαμε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των αρχών ε, υποδοχής και των ε, χωρών ε, και των αρχών της χώρας προέλευσης. τελικά όμως συμφώνησαν ότι διαφωνούν και αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδικασίες. Τώρα, ε, για την ώρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι φιλόδοξη προς την κατεύθυνση αυτή, διότι ε, σε όλες τις περιπτώσεις κοινών αποφάσεων υπάρχει πλέον υποχρεωτική διαμεσολάβηση εφόσον υπάρχει διαφωνία και όχι ξεχωριστέ αποφάσει και ξεχωριστέ διαδικασίε μεταξύ των δύο αρχών. Και αυτό για μας σημαίνει ότι όλες οι αποφάσει δεύτερου πυλώνα, ε, κεφάλαια, ρευστότητα είναι σημαντική αλλαγή. Εάν με ρωτάτε λοιπόν ε, για το κατά πόσο η πρόταση αυτή είναι κατάλληλη, ε, κάποια πράγματα θα τα γράφω διαφορετικά βέβαια, αλλά για την ώρα είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Διότι όπως είπα και νωρίτερα, αυτή του είδους η διακυβέρνηση έχει λειτουργήσει αρκετά καλά ε, σε κάποιους τομείς, αλλά ήταν λιγότερο αποτελεσματική σε άλλους. Ευχαριστώ. Έως τώρα κανείς δεν απάντησε στο ερώτημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο λύνει το θέμα ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου στην πρότασή τη. Ναι, πρώτα και το πρώτο μέρος του ερωτήματός σας ε, για την ε, διακυβέρνηση των αρχών και κατά πώς πρέπει να επεκταθεί. Για το εχειδίδιο του νέου κανόνα έχει λειτουργήσει καλά το σύστημα και αυτό φαίνεται και στην πρόταση. Εκεί όπου θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερους πόρους βέβαια σε επίπεδο αίσθημα είναι το θέμα της άμεσης ε, εποπτείας και της σύγκληση, της εποπτικής σύγκληση. Εκεί χρειαζόμαστε περισσότερες ε, αρμοδιότητες και θα πρέπει εκεί να δούμε και το θέμα, τα θέματα διακυβέρνησης. Ε, το υπάρχον μοντέλο που έχουμε ε, αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί αρκετά καλά. Θα ήταν ατυχές δηλαδή αν το αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης να οδηγήσει σε αλλαγή σε επίπεδο και όχι αλλαγή σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, διότι αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ε, ε, ταχύτητα με την οποία κινούνται, κινείται η οργάνωση. Ε, δηλαδή μπορεί να φαίνεται ότι ενισχύεται το σύστημα, αλλά εδώ ε, αυξάνουμε την διαδικασία, μεγαλώνουμε τη διαδικασία αντί να παίρνει την απόφαση ο πρόεδρος, δηλαδή περνάμε από το Συμβούλιο, ε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει αύξηση των εξουσιών, ε, αύξηση των πόρων, αλλά και ε, βελτίωση της διακυβέρνησης. Ευχαριστώ, συγγνώμη, Μπερές, δεν κυρία Μπερές, δεν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας, να θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του Προέδρου των Ευρωπαϊκών Αρχών, ο κεντρικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικός για μας το έχω πει εδώ και καιρό, αυξάνει την ε, λογοδοσία, αυξάνει την αξιοπιστία ε, της θέσης αυτής και θα πρέπει εκεί να γίνει μια προσαρμογή, για να είμαι ειλικρινής. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ECR έχει μόνο μία δυνατότητα να μιλήσει, οπότε θα σας κάνω μία ερώτηση στον καθένα. Προς την EBA η σχέση μεταξύ της ε, αρχής των τραπεζών και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού πώς ε, δουλεύει. Δεδομένου του ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην σύσταση αυτών των οργανισμών και συγκεκριμένα αν μπορούσατε να μας πείτε τι γίνεται σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θεωρείτε ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ σας και τι μπορεί να γίνει για την σχέση αυτή. Για τον κύριο Μπερναρντίνο Έχουμε κάποια θέματα εδώ με την, ε, με την προθεσμία του Φεβρουαρίου του 2018 και δεδομένου του ότι ακόμα δεν έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο οι τεχνικές προδιαγραφές σας, ε, θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε την προθεσμία μέχρι το Φεβρουάριο. Και πώς ενημερώνετε τα ενδιαφερόμενα μέρη για την τεχνική εργασία, δεδομένου του ότι πλησιάζει η προθεσμία. Και για την ΕΣΜΑ βέβαια δεν μπορώ να αφήσω τον κύριο Μαγιόρ να ξεφύγει έτσι, δεδομένου του ότι προσεχώς έχουμε, αρχές Ιανουαρίου δηλαδή, και την ημερομηνία εφαρμογή τη οδηγία με φοιτητή. Να σα ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν μπορείτε να μα ενημερώσετε για το πού βρίσκεστε σε σχέση με το νέο πληροφοριακό σύστημα που λέγεται Thirds και αν είναι σε καλό δρόμο. Και όσο πλησιάζει ο Ιανουάριος και ο κλάδος και ο τύπος ο σχετικός ε, σκέφτονται τα ζητήματα βλέπουμε πράγματα όπως ε, τα όρια των συνταγματικών συντημιών αλλά και το καθεστώς ε, των κινητών αξιών και βλέπουμε πως ε, πολύ μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μπορεί να περάσει σε κάποια γκρίζα ζώνη. Σας απασχολεί αυτό, πώς το αντιμετωπίζετε και αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κατάλληλες αντιδράσεις ε, από τις ανησυχίες οι οποίες από ό,τι αντιλαμβάνουμε υπάρχουν. Πολύ καλή ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι ακόμα πειραματιζόμαστε όσον αφορά την σχέση μας με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Δηλαδή εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι μια εποπτική αρχή όπως κάθε άλλη. Βεβαίως υπάρχουν εποπτικές αρχές ειδικά μετά την ε, απομάκρυνση, του, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι η αρχή η οποία θα υποπτεύει το 89% των ε, περισσιακών στοιχείων των ε, τραπεζών στο Ηνωμένο, στο, στην Ενωμένη Ευρώπη. Και βεβαίω η σχέση μα δεν είναι πολύ εύκολη για διάφορου λόγου. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια νομίζω πω ε, ήμασταν σε πολύ στενή συνεργασία. Από την αρχή είχαμε κοινό στόχο, ότι δηλαδή πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε σε διαφορετικά ζητήματα. Ο ξεκίνησε από τα κάτω, θα έλεγα, από τις εμπειρίες στο εθνικό επίπεδο και ανέπτυξαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα ενισχυθεί η ρυθμιστική πίεση ε, στις τράπεζες για να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Εμείς ε, εστιάσαμε περισσότερο στην αποτελεσματικότητα της αγοράς και την ανάγκη δημιουργίας μιας δευτερογενής, δευτερογενούς με συγχωρείτε, αγοράς ε, και δεδομένων, διαφάνειας κτλ. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι έχουμε τώρα εντολές από το Συμβούλιο να αναπτύξουμε καθημερινές γραμμές για τα κόκκινα δάνεια. Κάποιες από αυτές βασίζονται στην ε, εμπειρία και τις κατευθύνες γραμμές που είχε αναπτύξει ο νέος οπτικός μηχανισμός. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή να πηγαίνουμε από την ομοθεσία στις κατευθυντήριες γραμμές και μετά στην εποπτεία και την εφαρμογή, αλλά καμιά φορά γίνεται το αντίστροφο. Να πω ότι αντιλαμβάνομαι κάπως και τον ενίο μηχανισμό, γιατί πρέπει σήμερα να προχωρήσουν, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν πολλές διαφορετικές πρακτικές και πρέπει να αναπτύξουν κοινά κριτήρια για να επιτύχουν κάποια αποτελέσματα. Οπότε προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και οπωσδήποτε ο στόχος μας όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι κοινό. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά δεν περιμένουν τις κατευθύνες γραμμές σας. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την ερώτηση. Πράγματι για την εφαρμογή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει αυτά τα χρόνια για να μπορέσουμε να δώσουμε την συμβουλή μας στην ε, Κομισιόν. Επίση, ε, έχουμε μπλακεί με τους συμμετέχοντες στην αγορά και στη δημόσια διαβούλευση και σε άτυπες συναντήσεις, ε, έρωτο αποκρίσεις. Υπ' αυτήν την έννοια κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε σε επαφή με τους συμμετέχοντες ε, στην αγορά, οπότε δεν υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις. Όσον αφορά λοιπόν ε, την εφαρμογή τέτοιων αλλαγών, πάντα υπάρχει το θέμα των ε, δυνατοτήτων της πληροφορικής για να γίνουν εγκαίρως αυτές οι αλλαγές. Και εκεί πέρα ακριβώ πρέπει να αντιληφθούμε το εάν ολόκληρη η αγορά στην Ευρώπη θα μπορεί να λειτουργήσει τον Φεβρουάριο του 2018. Μα ακούμε κάποια μηνύματα από εδώ και από εκεί και για να είμαι ειλικρινής μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα, αλλά αυτό είναι και ένα μάθημα για το μέλλον. Πρέπει να δώσουμε νομίζω λίγο περισσότερο χρόνο όσον αφορά τη στιγμή μεταξύ της οποίας ε, καταλήγουμε στο ρυθμιστικό πλαίσιο και της πραγματικής εφαρμογής, γιατί υπάρχει και το θέμα της ε, πρακτικής εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων. Ευχαριστώ για τα ερωτήματα. Να σας ενημερώσω καταρχήν ε, για το FERTS, το οποίο είναι πρόσφατο ακρόνιμο, είναι ενδιαφέρον ε, project. Πρόκειται για μια εθνική υποχρέωση η οποία πλέον έχει ανατεθεί στην ΕΣΜΑ προς τα πάνω δηλαδή. Ε, είναι και μια πρόταση της Επιτροπής όπου κάποια από τα δεδομένα αυτά και τις σχετικές, σχετικές ευθύνε ε, δίνονται πλέον στην ΕΣΜΑ. Αυτό ενισχύει το σύστημα. Έτσι δεν χρειάζεται να περάσουμε από αυτήν την χρονική περίοδο που πρέπει να περιμένουμε να φτάσει το project στο επίπεδο ΕΣΜΑ. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε βέβαια ότι θα λειτουργήσει αυτό. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί σωστά και θα φέρει αποτελέσματα από τον Ιανουάριο του 2018 και μετά. Ε, πρέπει να σας ενημερώσω ότι εμείς συνδέσαμε με πάνω από 300 διαφορετικούς ε, ε, διαφορετικές χρηματαγορές ε, τα στοιχεία αυτά. Τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησε η διαδικασία και ε, λογικά θα πρέπει να αρχίσουμε να συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά την, από τον Ιανουάριο του 2018. Θα είμαστε έτοιμοι. Και το 2018, ανάλογα και με τον τύπο των ε, χρηματοοικονομικών μέσων που θα έχουμε στη διάθεσή μας ε, θα δημοσιεύουμε ε, τα στοιχεία αυτά εντός 2018. Βεβαίως τον Ιανουάριο 2018, 2018 το αμύφι θα πρέπει να, αρχίσει να λειτουργεί ήδη, οπότε έχουμε ήδη δημοσιεύσει κάποια από τα με, κάποιους μεταβατικούς υπολογισμούς και ελπίζουμε όλα αυτά να μπορέσουν να δημοσιευθούν πριν το τέλος του έτους. Είμαι αρκετά αισιόδοξο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του FITS, όμως πρέπει να πω ότι εξαρτάται και από την ποιότητα των δεδομένων που θα λαμβάνουμε από τις χρηματαγορές και βεβαίως συνεργαζόμαστε με τα trading venues αυτά, αλλά χρειάζεται και δική του συνεργασία για να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία και η διαφάνεια θα διέπουν αυτό το σύστημα και θα είναι ποιοτικά τα στοιχεία. Ε, η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι είμαστε σε καλό δρόμο πάντως. Ό,τι αφορά το καθεστώς SI, ε, βεβαίως ε, είναι ένα καθεστώς το οποίο οδηγεί σε λιγότερη διαφάνεια, ε, ρυθμιζόμενες αγορές, MTS. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι το καθεστώς SI δεν θα χρησιμοποιηθεί για να παρακάμψει κανείς ε, τους στόχους του MIFID 2. Έχουμε ήδη τρεις δράσεις από κοινού με την εικόν. Έχουμε κλείσει ένα από τα κενά που υπήρχε. Ε, είναι η πρωτοβουλία του Μάρκους Φέρμπερ που έχει να κάνει με τον κίνδυνο ε, ενός κενού το οποίο λύθηκε μέσω μιας κραξιότητας πράξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε τα SI ε, να μην συνδέονται μεταξύ τους και να μπορούν να κάνουν αυτή την παράκαμψη. Πρόσφατα είχαμε ένα Q&A για τα SI, τα οποία ε, θα πρέπει να δημοσιεύουν τις πληροφορίες ε, όσο γρήγορα, με την ίδια ταχύτητα με τις χρηματαγορές. Ε, επίσης, θέλουμε να δούμε κατά πόσο το καθεστώς για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που να χρησιμοποιηθεί και για τα ζητήματα διαφάνειας σε επίπεδο SIs. Ευχαριστώ. Ο Φίλιπ Λαμπέρτς έχει τον λόγο τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Έχω τρία ερωτήματα ε, και στους τρεις σας και μετά έχω και μία για τον κύριο Ενδρία. Πρώτα για τον Brexit. Οι πόροι που έχει στη διάθεσή σας αρκούν για να εξασφαλίσετε την σωστή εποπτεία αυτών που θα κάνει το Ρωμένο Βασίλειο, διότι οι νομοθεσίες μετά τον Brexit θα αποκλίνουν. Ε, είναι σημαντικό όμως εσείς ε, να μπορέσετε να παρακολουθείτε, να υποπτεύετε τις εξελίξεις, ιδιαίτερα αν υπάρξει κάποια ισοδυναμία. Πιστεύετε ότι έχετε του επαρκεί πόρου. Δεύτερον, πάντα για του πόρου. Θεωρείτε ότι το νέο καθεστώ χρηματοδότηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι καλό. Δίνεται μεγαλύτερο έμφαση στα τέλη σε ό,τι αφορά την εποπτεία. Μήπω εδώ υποκύψουν και συγκρούσει συμφερόντων. Ε, Επίση, θα είναι επαρκή τα χρήματα αυτά, τα τέλη αυτά. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε η Περβάνο προηγουμένω για τη διακυβέρνηση, έχουμε δει ότι τα RTS ε, ε, έχουν κολλήσει εκεί στην ΕΠΑ. Στο άρθρο 124 ε, δίνονται κάποιες δυνατότητες ε, και εκεί δεν μπορεί να υπάρξει έγκριση όμως. Πιστεύετε ότι το νέο καθεστώς, η νέα κυβέρνηση θα σας επιτρέψει να μπορεί να παίρνετε αποφάσεις πιο εύκολα. Εμείς πάντα ήμασταν υπέρ να έχετε εσείς κάποιες εξουσίες ως πρόεδροι ε, δεν φαίνεται βεβαίω να συμβαίνει αυτό την πρόσθεση της Κομισιόν. Ε, κύριε Ένρια, έχετε ένα δύσκολο έργο, και τρει έχετε δύσκολο έργο βέβαια, αλλά ε, αυτή τη στιγμή είστε στον Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε δεν θα γνωρίζετε ότι εκεί λαμβάνει η χώρα μια συζήτηση. ο Τζον Φίγκερ, παραδείγματο χάρη, αναφέρεται συχνά στην ανάγκη να είναι οι ψηλότερα arm funds που θα απλοποιεί πολύ την ρύθμιση βέβαια διότι εάν έχουμε 20% μόχλευση τότε μπορεί να υπάρχει ένα μεγάλο μέρος που να αποκλείεται. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τη γνώμη σας. Μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό έτσι ώστε όλες ε, οι τράπεζες να είναι πιο ανθεκτικές. Λοιπόν πρώτα η ΕΣΜΑ. Τρία λεπτά συνολικά, έτσι. Θα είμαι σύντομος ε, για το θέμα των πόρων. Ήδη στα αρχικά μου σχόλια σας είπα ότι κάποια στοιχεία για το ΜΥΦΙΛ 2 παραδείγματος χάρη ε, έπρεπε να υπάρξει μια μεταβατική φάση. Το ιδανικό θα ήταν βεβαίως ε, να έχουμε το κατάλληλο μέγεθος πόρων για να αντιδράσουμε. Τώρα για το Brexit, όχι μόνο των τον Βασιλείο, αλλά και τώρα, από τώρα, ετοιμαζόμαστε γι' αυτό και ήδη αυτό μας απασχολεί, απασχολεί πολύ χρόνο και πόρους. Εάν θέλουμε να, κάνουμε μια, να έχουμε μια αξιόπιστη αξιολόγηση των κινδύνων ε, που ελοχεύουν στα πλαίσια του Brexit, χρειαζόμαστε πολλούς πόρους. Και εδώ έχουμε αφαιρέσει πόρους από άλλες, άλλα θύματα προτεραιότητων στα ότι Είναι σημαντικό βέβαια στο θέμα του Brexit, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι εδώ. Αλλά ετησίως δημοσιεύουμε το πρόγραμμα εργασιών και εκεί φαίνεται ποια είναι, ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φέρουμε σε πέρα επειδή δεν έχουμε επαρκεί πόρου. Και εδώ πρέπει να είμαι διαφανή. Υπάρχουν και νομικέ υποχρεώσει. Κάποιε υποχρεώσει ε, σχετικά με τι βάσει δεδομένων που προέρχονται από του νομοθέτε. Εμεί έχουμε πει ανοιχτά ότι δεν μπορούμε να αντιποκριθούμε στι υποχρεώσει αυτέ γιατί δεν έχουμε του πόρου. Ε, με αυτή την έννοια λοιπόν χρειαζόμαστε πιο πολλούς πόρους. Βεβαίως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ δηλαδή με τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται εκεί. Ευχαριστώ. Ναι, σε σχέση με το Brexit, ήδη για την ισοδυναμία, ε, ο πόρος, οι πόροι που έχουμε στη θέση μας ε, για να εποπτεύουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις εξελίξεις στις χώρες όπου ήδη παίρνουν τα αποφάσεις αδυναμίας είναι ε, οι πόροι αυτοί. Τώρα, αν προκύψουν προβλήμα με το Μένο Βασίλειο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Θέλω όμω να επιζήσω την προσοχή σα σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι έω τώρα, ε, σε ό,τι αφορά την ισοδυναμία, εμεί πάντα επικεντρωνόμασταν ε, στην ε, εποπτεία τη εξέλιξη τη ρύθμιση. Πρέπει όμω να εποπτεύσουμε την εφαρμογή της ρύθμισης, την εφαρμογή του κανονισμού, διότι εκεί προκύπτουν οι διαφορές. Ε, όπως σημαίνει και στην Ευρώπη, στο έργο που γίνει σε επίπεδο σύγκληση τη εποπτεία, πρέπει να αυξηθούν τα καθήκοντά μα ε, όταν παίρνουν αποφάσει ισοδυναμία, δηλαδή να μπορούμε να εποπτεύουμε την εφαρμογή του καθεστώτος. Ε, εκεί ε, προκύπτουν οι μεγάλε διαφορέ. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν έχουμε πόρου γι' αυτό. Και στην πρόσθεση τη Κομισιόν, ε, τουλάχιστον για μας, ε, δεν αρκούν οι πόροι που προτείνονται για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το σκέλος της εφαρμογής ε, για τη χρηματοδότηση. Βεβαίως ε, είμαστε υπέρ των τελών. Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι δεν έχουμε το καλύτερο δυνατό σύστημα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε βεβαίως ότι στη δικασία αποφάσεων που παίρνουμε για τα τέλη τα οποία θα συλλέγουμε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Διότι ζούμε στην Ευρώπη, έτσι. Οι αποφάσει θα παρθούν από τι δημοσιονομικέ αρχέ, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο τελικά. Είναι σημαντικό όμω αυτά να τα συνδυάσουμε με την ανεξαρτησία. Όπω προβλέπεται στην, αρχή, στην πρόταση τη Κομισιόν αυτή τη στιγμή. Διότι δεν υπάρχει καμιά παρέμβαση σε ό,τι αφορά τι αποφάσει που θα παίρνονται σε επίπεδο αρχών αλλά και σε ό,τι αφορά τα πρόγραμμα εργασιών των αρχών μας. Αυτό πρέπει να παραμείνει, διότι είναι πολύ σημαντικό, ε, συνδέεται με την εξέλιξη ε, της χρηματοδότησης ε, και με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας. Ναι, δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Η ισοδυναμία, βεβαίως, ε, ε, η υποπτία της ισοδυναμίας σημαίνει ότι χρειαστούμε, χρειαστούμε πολλούς περισσότερους πόρους. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύγκρουση συμφερόντων, ε, ακούστε, υπάρχουν πολλές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές που χρηματοδοτούνται από τον κλάδο. Ε, μπορούμε να προστατεύσουμε την αρχή από τη σύγκρουση συμφερόντων, νομίζω. Τώρα για τη διακυβέρνηση και το RTS, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί πάντα να εκδώσει το RTS και με το παρόν σύστημα. Εάν δηλαδή δεν παραδώσουμε εμεί το RTS εντό τη προθεσμία, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει. Εμεί έχουμε κάνει το παρασκευαστικό έργο, δηλαδή είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Εάν θέλετε τώρα ο πρόεδρο ε, να μπορεί να ψηφίσει κατά να, ψηφίσει με κάποια ειδική ψηφοφορία και να αποφασίσει, εντάξει, εδώ μπλέκονται και προσωπικά μου συμφέροντα, αλλά ε, είναι σωστό σίγουρα να υπάρχει περισσότερη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, για το θέμα του Βίκερς, ακούστε, είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε τους δύο πόλους ε, ε, τη συζήτηση για τα κεφάλαια, κατά πόσο τα κεφάλαια είναι τα κατάλληλα στις τράπεζες. Κάποιοι λένε ότι είναι πολύ ψηλά τα κεφάλαια, από τις τράπεζες, ότι αυτό παρεμποδίζει τη χρηματοδότηση της ε, οικονομίας. Από την άλλη υπάρχει ε, ένα σημαντικό μέρος ακαδημαϊκό, που λέει ότι είναι πολύ χαμηλό και ότι πρέπει να έχουμε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα κεφαλαίων. Ε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί, ε, τελικά έχουμε ένα υψηλό επίπεδο απαιτήσεων κεφαλαίων, αλλά διαχειρίσιμο. Και βεβαίω ε, αυτό που είπατε εσεί. για τους άλλους, για τους άλλους τύπους κεφαλαίων, δηλαδή κάποια εργαλεία, κάποια μέσα που μπορεί να αυτή τη στιγμή είναι νεκρά, αλλά μπορούν να μετατραπούν σε κεφάλαια. Αν μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί οι μηχανισμοί, ε, νομίζω ότι θα είμαστε αρκετά καλά σε επίπεδο κεφαλαίων. Εάν δούμε ότι στην εφαρμογή της σύγκλησης, ε, στην εφαρμογή αυτών των μέσων τα πράγματα δεν λειτουργούν, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι παρκές το επίπεδο κεφαλαίων. Έτσι το βλέπω εγώ. Eh, να επιστρέψω λίγο στα MPL και τους δείκτες οι οποίοι χειροτέρευσαν σύμφωνα με αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς είπατε ότι το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να καταθέσει σύντομα τις κατευθυντήριες γραμμές, αλλά επί της ουσίας διαρωτώ με η εντολή αυτή είχε σαν στόχο να δημοσιεύσετε το 2008 τις ε, κατευθυντήριες γραμμές της ε, τραπεζικής αρχής. Για ποιο λόγο ε, κυκλοφόρησαν τα στοιχεία αυτά ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, στοιχεία τα οποία δημιούργησαν κάποιο πανικό στις αγορές. Και τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με τις πραγματικές προθέσεις αυτών οι οποίοι τα κυκλοφόρησαν. Αυτό οδήγησε σε πάρα πολλές πωλήσει στην Ιταλία. Γενικά θα πρέπει να δούμε αν κάποιες, κάποιες οντότητες ισχυρές, τρεις ή τέσσερις είναι που διαχειρίζονται τα MPLs, είχαν κάτι να κερδίσουν από αυτό. Σε άλλες χώρες στο παρελθόν ε, δόθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν λίγο το θέμα αυτό. Στην Ιταλία όμως είμαστε πάρα πολύ πίσω και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο επίπεδο στρέβλωσης της πιστοτικής των τραπεζικών αγορών. Συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσετε να μας εξηγήσετε αν αυτή η σημαντική στρέβλωση στις πιστοτικές αγορές ε, έχει σχέση και με τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν αυτά τα στοιχεία. Τώρα για το τρίτο επίπεδο θα ήθελα διαβεβαιώσεις από πλευρά σας να μας πείτε τα επόμενα stress test αν θα συνοδεύονται και από πραγματικές ε, διαδικασίες αξιολόγησης. γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία των τραπεζών, ε, τα οποία από ό,τι λένε κάποιοι πολύ σοβαροί αναλυτές, δεν λαμβάνονται υπόψη καθόλου από την Ευρωπαϊκή Αρχή. Ευχαριστώ κύριε Βάλλη. να προσπαθήσω να εξηγήσω λίγο πώς ε, εμείς συνδεόμεθα σε επίπεδο κατευθυντηρίων γραμμών με το SSM. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από το SSM για το πώς αυτή τη στιγμή σε καθημερινή βάση μπορεί να διαχειρίζεται κανείς το χαρτιφυλάκιο των MPLs. και μάλιστα πολλά από τα στοιχεία αυτά προήλθαν από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας η οποία έχει τεράστια εμπειρία στα πλαίσια της επιτυχούς κατά τα άλλα διαχείρισης των χαρτοφυλακίων αυτών. Στα πλαίσια λοιπόν των συζητήσεων του θέματος αυτού, αποφασίσαμε ότι επί τη βάση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών θα μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε ορισμένα στοιχεία, να διευρύνουμε αν θέλετε το πεδίο κυκλοφορίας των στοιχείων αυτών με πρωτοβουλία του SSM. Εμείς λοιπόν βασιζόμαστε και στις δικές μας, θα βασιστούμε στις δικές μας κατευθυντήριες γραμμές, στις προσπάθειες τις οποίες έχει ήδη κάνει ο SSM. Έχει κυκλοφορήσει και ένα παράρτημα ή μία προσθήκη αν θέλετε σε αυτές τις πρώτες κατευθυντήριες γραμμές που ασχολείται με τα νέες αρροές των ε, κόκκινων δανείων και έχει σαν στόχο να μην δημιουργηθεί μια νέα σόρευση αν θέλετε, τέτοιου είδους δανείων, ενώ προσπαθούμε, προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τα παλαιότερα. Και γι' αυτό λοιπόν και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμείς λαμβάνουμε υπόψη και θα το συζητήσουμε φυσικά και με τον SSM. Η βασική αρχή λοιπόν που οδήγησε στην κυκλοφορία των στοιχείων αυτών δεν είναι λανθασμένη. Από την άλλη το θέμα είναι πώς χρησιμοποιούνται στην πρακτική. Ε, υποτίθεται ότι η τραπεζική αγορά στις Ηνωμένε Πολιτείες αντιμετώπισε το θέμα των κόκκινων δανείων με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να πάρουμε στοιχεία από το SSC που προβλέπει ότι στο εξάμεινο μη εξυπηρέτησης πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τα θέματα λοιπόν του επόμενου stress test θα δημοσιεύσουμε κάποια πρώτα στοιχεία τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου και θα είναι έτσι και αλλιώ στο ε, τμήμα ε, των κατευθυντήριων γραμμών. Να θυμίσω ότι τα stress tests δεν είναι στοιχείο αξιολόγησης. Ε, αν τυχόν οι, εξ, αξιολογήσεις βασίζονται αποκλειστικά πάνω στα ευρήματα αυτών των τεστ, νομίζω ότι αυτό θα είναι ανεπαρκές. Ματό. Όχι. Μονό. Συγγνώμη. Μονό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γκαμπριέλ Μάτο. Να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές για την εξαιρετική τους παρουσίαση. Να πω στον κύριο Ενρία, θα συμφωνήσετε μαζί του, μαζί μου συγγνώμη, ότι ε, θα πρέπει οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές να αντικατοπτρίζουν, ε, ε, θα έλεγα, μια σταθερή κατάσταση γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια στάθεια στις ε, τραπεζικές αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία μπορεί να επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το θέμα είναι να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα θέματα που άπτονται των τρίτων χωρών. Ε, ποια είναι τα προγράμματα και ποιες, ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχετε για την αναγνώριση την λεγόμενη των τρίτων χωρών. Και τώρα για τις τράπεζες με πολλαπλά σημεία εισόδου, multiple point of entries. Πώς ε, μπορούμε εμείς ε, να δούμε ε, τις διαφορές στη διαχείριση και στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων single point of entry ενός μοναδικού σημείου εισόδου και πολλαπλών σημείων εισόδου. Τώρα, για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από πλευράς ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες. Ε, θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος αυτού του τύπου των υπηρεσιών και υπάρχουν κάποιοι ειδικοί λόγοι που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση του ελέγχου της άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων. Και στα πλαίσια της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών τι γίνεται για μονάδες οι οποίες δημιουργούνται σε μία χώρα με μοναδικό στόχο να δραστηριοποιηθούν σε άλλη χώρα. Συνειδητοποιώ λοιπόν το επίπεδο της ερώτησης νομίζω και περιμένω μια απάντηση από πλευρά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, για την ισοδυναμία τρίτων χωρών μας απασχολεί αυτή τη στιγμή έχουμε πράγματι μείνει πίσω. Ε, συχνά λαμβάνω επιστολές από διοικητές ε, υποπτικών συμβουλίων και λένε να επιταχύνουμε στην αναγνώριση της ισοδυναμίας ε, των δικαιοδοσιών γιατί έχει μεγάλη, έχουν μεγάλη παρουσία εκεί οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Και βέβαια έχει σημασία για τη χρηματοδότηση των οικονομιών τους. Όπως σωστά λέτε είναι ζήτημα πόρων έχουμε ένα άτομο. Είχαμε ένα άτομο που έκανε αυτή τη δουλειά, έφυγε και δεν ε, μπορέσαμε να τον αντικαταστήσουμε εδώ και ένα έτος. Ε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε πάλι προσλήψεις. Ξεκινήσαμε νέες δύο, δύο με συγχωρείτε, νέες διαδικασίες ισοδυναμίας στην Παρασκευή που μας πέρασαν. και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα γιατί η ισοδυναμία τρίτων χωρών πρέπει να αναγνωριστεί μέχρι το τέλος του επόμενου έτους για να αποφύγουμε το ότι το κρατικό χρέος αυτών χωρών θα πέσει σε μη προτιμησιακή μεταχείριση όσον αφορά τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις των τραπεζών. Τώρα για τα διάφορα μοντέλα MP, SP κτλ. Εμείς ως εποπτικές αρχές θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι όσον αφορά τις επιλογές των τραπεζών ε, είτε μιλάμε για διασυνοριακή, σε διασυνοριακή βασικά ένα ή πολλαπλά σημεία ε, εισόδου. Θα πρέπει απλά να υπάρχει ένα σύστημα διάσωσης το οποίο θα λειτουργεί οποιοδήποτε μοντέλο και αν επιλέξουν να ακολουθήσουν οι τράπεζες σε περίπτωση κρίσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Η σημαντικό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι τώρα με την φερικαιότητα 2 και τις ε, απαιτήσει ε, αναφορών που έχουμε αυτή τη στιγμή με πάνω από 3.000 εταιρείε που στέλνουν πληροφορίες σε εθνικές αρχές και μετά σε εμάς έχουμε πολύ περισσότερες ε, πληροφορίες για το πώς υπάρχουν αυτές οι ροές οι Γιατί στο παρελθόν, σε περιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών, η κάθε υποπτική αρχή έπρεπε να δώσει κάποιε πληροφορίε στις σχετικέ εταιρείε και δεν γινόταν αυτό τι περισσότερε. φορές. Τώρα όμως υπάρχει η ΕΙΟΠΑ σε μια κεντρική θέση και εμείς θέλουμε για πρώτη φορά στις εθνικέ αρχέ, την πληροφορία του τι γίνεται, ποιε συναλλαγέ γίνονται σε κάθε Και βεβαίως και με τον αυξανόμενο ρόλο μας, καθώ κοιτάμε και από υποπτική σκοπιά το τι συμβαίνει στην αγορά, ε, έχουμε δει, όπως είπα, κάποιες διασυνοριακές καταστάσεις όπου είχαμε κάποιες χρεοκοπίες. Και βεβαίως αυτό μας κινητοποίησε και σχηματίσαμε αυτέ τις πλατφόρμες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα στην παρέμβασή μου, να φροντίσουμε ότι θα γνωρίζουμε αυτές τις περιπτώσεις πολύ πριν φτάσουμε στην αφαιρεγγιότητα. Αλλιώς ε, θα έχουμε τον ρόλο της συντονίζουσας εποπτικής αρχής, αλλά δεν θα τα γνωρίζουμε αυτά πριν να είναι πολύ αργά. αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωμένε οι εθνικές αρχές από τον κανονισμό να μας ενημερώνουν όταν υπάρχει κάτι το οποίο πάει στραβά και έχει διασυνοριακή διάσταση. Κάτι άλλο το οποίο δεν είναι ιδανικό θα έλεγα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές διαστάσεις, δηλαδή το ίδιο άτομο όταν πηγαίνει από την ε, μία χώρα θεωρείται ικανός και κατάλληλος σε μια χώρα στην οποία πηγαίνει και όχι στην χώρα από την οποία ξεκίνησε. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες ασυνέπειες και κάποια περίεργα μοντέλα. Τώρα λοιπόν γνωρίζουμε αυτές τις ε, καταστάσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη έντολη για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή η οποία θα εξετάζει ακριβώς όλους τους ασφαλισμένους στην Ευρώπη ειδικά όταν υπάρχει διασυνοριακή διάσταση. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω και εγώ μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις. Μία προ τον κύριο Νερία, μία προ τον πρόεδρο τη ΕΣΜΑ. Μιλήσατε μόλις για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπου εγώ βλέπω δύο διαφορετικά προβλήματα. Το ένα είναι νομικό, μεθοδολογικό και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία, κατευθυντήριε γραμμές και ρυθμιστικές αρχές. Από ό,τι φαίνεται δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και θα πρέπει και εμείς ως νομοθέτες να δούμε την νομική βάση, η οποία θεωρώ ότι δεν ε, στέκει ιδιαίτερα. Βεβαίω αυτό δεν είναι ερώτηση, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η σχετική οδηγία για κεφαλαϊκές απαιτήσει θα γίνει το μήνυμα. Κοιτάξτε. Ε, Ετέθη το ζήτημα της ροής των ε, νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, και κάποιου αποθέματος. Οπότε ένα παλαιό δάνειο, παραδείγματος χάρη, το οποίο γίνεται μη εξυπηρετούμενο. Και μετά υπάρχει εδώ πέρα μια περίεργη διατύπωση ε, στο δελτίο τύπου, όπου μιλάτε λέτε κάτι για το απόθεμα κάτι το οποίο δημιουργεί κάποιες αναταράξεις στην αγορά. Θεωρείτε λοιπόν ότι οικονομικά έχει νόημα να χρησιμοποιούμε την ίδια προσέγγιση για το απόθεμα και για την ροή, καθώς δεν θέλουμε να διαταράξουμε την αγορά αυτή, η οποία σιγά σιγά ανακάμπτει και βλέπουμε μια αύξηση τιμών και πλησιάζει η τιμή της αγοράς λίγο περισσότερο στην πραγματική τιμή γιατί όποιος ε, θεωρεί ότι θα πρέπει να δούμε διαφορετικά το απόθεμα θα σκεφτόταν κάποια διαφορετικά μέτρα και όχι απλά μια γραμμή σε μια διαβούλευση γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύσει. Η δεύτερη σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Μαγιόρ για τα νέα καθήκοντα που σας δίνονται για τα CCP. Ε, γιατί τώρα μελετάμε μία πρόταση, έχουμε και ένα εκτελεστικό ε, συμβούλιο και μια εκτελεστική συνέλευση και μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς βλέπετε να επιδρούν όλοι αυτοί οι φορείς. Γιατί έχουμε το Γενικό Συμβούλιο τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ, τον πρόεδρο της συνέλευσης, τον εκτελεστικό διευθυντή της ΕΣΜΑ, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν συμφωνεί εκτελεστική συνέλευση και μετά υπάρχουν οι δεσμευτικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειλικρινά δηλαδή το βρίσκω λίγο περίπλοκο εκ πρώτης όψεως, αλλά ίσως κάνει λάθος. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μας πείτε. Ο Ανδρέα πρώτος. Ε, thank you, thank you, ε, Roberto. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, γιατί θα απαντήσω έτσι και σε ένα τμήμα της ερώτησης βάλει το οποίο δεν κάλυψα. Τώρα, στόκ από τη μία απέναντι στις ροές από την άλλη. Τώρα, η προσπάθεια αποτροπής μιας νέας σώρευσης μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι κάτι το οποίο αν δεν το πετύχουμε ε, θα οδηγηθούν οι τράπεζες σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα το αποτρέψουμε. Εξακολουθούμε να έχουμε ένα σύνολο βέβαια μη εξυπηρετούμενων δανείων και σε αυτό τον τομέα η δική μας σύσταση ε, είναι να ε, αυξηθεί η εποπτική πίεση και αυτή τη στιγμή αυξηθεί η πίεση αυτή να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε ε, το push με το pull, δηλαδή κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τις ισορροπίες της ίδιας της αγοράς, να συνεργαστούμε με ε, επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων και ενεργών στοιχείων, Υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες ε, ε, κυριαρχούν στην αγορά. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται αυτού του είδους ε, τα δάνεια και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να βρούμε νέους επενδυτές και να μπορέσουμε έτσι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με καλύτερο τρόπο. Η πίεση λοιπόν η εποπτική θα πρέπει να σταθμιστεί και σε σχέση με την ικανότητα απορρόφησης της αγοράς. Να πω επίσης ότι εγώ ε, την προσθήκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν την ερμηνεύω σαν μια πρόταση αυτόματης ε, παράτασης της πρότασης η οποία υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ότι κάνουμε για τα στόκ των δανείων το ίδιο να κάνουμε και για τα νέα δάνεια τα οποία εισέρχονται. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να εγγυηθούμε είναι η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια ε, των, ε, των αγορών δευτέρου επίπεδου. Να πω πρώτα ότι υποστηρίζω σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της, σε περιπτώσει. Οι υποδομέ είναι ακριβώς ένα τομέα όπου μπορεί να υπάρξουν ωφέλη εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό αυτών των υποδομών, να μπορούμε να κάνουμε κλίμακα να μπορούμε να εκπαιδευτούμε την πραγματογνωμοσύνη που έχει συγκεντρωθεί, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι 10 με 15 ο αριθμός. Ε, δεν μπορούν οι εθνικές και εθνικές αρχές, να το διαχειριστούν αυτό. Ε, είναι, είναι πολλά τα επιχειρήματα και μια κεντρική εποπτεία. Επίσης η απάντηση από το Συμβούλιο των Εποπτικών Αρχών ε, ήταν ακριβώς αυτή, να υπάρξει συγκεντρωτισμός σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εποπτεία. Οπότε συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, ε, βεβαίως σε μια σειρά από η πρόταση είναι περίπλοκη, είναι αρκετά περίπλοκη. Και είναι σημαντικό να έχουμε ένα καθεστώς διακυβέρνηση και δίπλη λήψη αποφάσεων που όπου θα είναι σαφές το ποιο αποφασίζει και να παίρνουν οι αποφάσει έγκαιρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που πρέπει να βγουν από την πρόταση. Πρώτον, το γεγονό ότι για μια σειρά αποφάσει όχι μόνο η υποστήριξη τη κλειστική εξουσία χρειάζεται, αλλά, αλλά και από την Κεντρική Τράπεζα ε, έκδοση. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί έγκριση. Εκεί τι θα γίνει αν δεν συμφωνήσουν όμω. Διότι δεν υπάρχει διαμεσολάβηση και δεν υπάρχει λύση. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Μια δυνατότητα είναι να υπάρξει μια δια... Ε, διαβούλευσης. Ε, μια άλλη δυνατότητα είναι η κεντρική τράπεζα να είναι αυτή που θα αποφασίζει. Ε, δεν είναι πάντως καλό να έχουμε παράλληλα δύο συστήματα λήψη αποφάσεων χωρίς να είναι σαφές το τι συμβαίνει όταν αποκλίνουν ε, στις εκτιμήσεις τους. Το άλλο θέμα είναι ο συνδυασμός μεταξύ της executive session και του ε, Συμβουλίου της Υποπτικής Αρχής. Πρώτα απ' όλα, όσο έχει πρόταση, ε, η Εκλεστική Επιτροπή θα έχει μια διαφορετική στρατηγική, διαφορετική εξωτερική εκπροσώπηση και κυρίως θα χρησιμοποιεί τους πόρους της ΕΣΜΑ, αλλά δεν θα έχουμε ε, μια, ένα κοινό σώμα ψηλά στην πυραμίδα της οργάνωσης θα παίρνουν αποφάσει από το εκτελεστικό αυτό όργανο, θα δίνει παραδείγματο χάρη, θα δίνει, παραδείγματος χάρη συμβουλές στις εθνικές εποπτικές αρχές, όμως το ε, συμβούλιο είναι αυτό που θα είναι υπεύθυνο για τα Q&A, για τα stress test κτλ. Και εκεί μπορεί να υπάρξει ασυνέπεια, μπορεί να υπάρξει απόκληση στην λήψη αποφάσεων και αυτό δεν θα βοηθήσει. Έτσι και λοιπόν κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ευθυγραμμίσουμε αυτά τα όργανα όσο γίνεται περισσότερο. Η ΕΣΑ στην πρόταση αναθεώρησης ε, είναι ένας τρόπος αυτός ε, για να αποφύγουμε τις επικαλύψεις μεταξύ της Executive Station και του Executive Board. Ε, βλέπετε ότι βεβαίως ότι είναι σχεδόν ίδια η συμμετοχή. θα πρέπει να προφροντίσουμε μάλλον να είναι οι ίδιοι εκπρόσωποι και στα δύο όργανα έτσι ώστε να παίρνονται οι ίδιες αποφάσεις από τα όργανα ουσιαστικά. Ευχαριστώ θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη συνέπεια, διότι είναι σημαντικό αυτό και σε επίπεδο νομοθετική διαδικασία. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο περίπλοκο, αν θέλετε. Και τώρα το λόγο έχει η Ντανούτα, η συγγήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ο Ρομπέρτο μου έκλεψε το ερώτημα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να μπορέσει η διαδικασία λήψη αποφάσεων να είναι όσο γίνεται πιο συνεπή. Είναι σημαντικό αυτό. Οπότε έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα προς τον κύριο Αντριά για τον Brexit. Όλες οι συναντήσεις που είχαμε με τον χρηματοοικονομικό κόσμο μας λένε ότι προετοιμάζονται για το σκληρό Brexit, το hard Brexit, αυτό το σενάριο. Φαντάζομαι ότι και εσείς ε, είστε υποχρεωμένοι να λάβετε υπόψη σας και αυτή τη δυνατότητα. Ε, ότι, να έχουν, ότι μπορεί να έχουμε δηλαδή και σκληρό Brexit παρότι βεβαίως δεν το θέλει κανείς. Ε, πολλά όμω από τα θέματα, αναφέρθηκα στον κλάδο, αλλά πολλά, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Brexit είναι στα χέρια σας. Ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό που έχετε κάνει ω τώρα με γραμμέ γραμμές και όλα αυτά τα, ε, όλες τις που έχετε πάρει. Αλλά το ερώτημά μου έχει να κάνει με το εξή. Όλοι θέλουμε να αποφύγουμε ε, να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει ένα κενό κέλυφος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Υπάρχει το θέμα τη τρίτη διακυβέρνηση, υπάρχει το θέμα τη ανάλυση κινδύνου, και της αξιολόγησης τη διαχείριση κινδύνου στα πλαίσια του Brexit. Ε, η ΕΜΠΑ έχει κάνει κάποια ανάλυση ε, σε ό,τι αφορά το back-to-back -back model στην περίπτωση του Brexit. Ε, μπορεί να έχουμε εδώ ένα κενό κέλυφο, αλλά, αλλά αν το προετοιμάσουμε καλά μπορεί να είναι και μια λύση για την κατάσταση μετά το Brexit. Έχετε κάνει κάποια ανάλυση προ την κατεύθυνση αυτή, το έχετε σκεφτεί. Ε, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να γίνει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά ενδεχομένω και λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, ε, σύντομα θα δημοσιεύσουμε μια γνωμάτευση που θα αναφέρει και το κεφάλαιο για την εσωτερική διακυβέρνηση, για το outsourcing, το back-to-back -back και αυτές τις μεταβιβάσεις εντός ε, της ομάδας. Ε, είναι μια κλειδιά αυτά, τα οποία γίνονται όλο και πιο επίκαιρα. Ε, υπάρχουν πρακτικές λύσεις. Οι διεθνεί ε, τράπεζε επενδύσει βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια του back-to-back για να μπορέσουμε να μειώσουμε και να συγκεντρώσουμε τον κίνδυνο. Ε, δεν θέλουμε βεβαίω του μηχανισμού να του διαταράξουμε. Από την άλλη, θέλουμε να αποφύγουμε το κενό κέλυφος, τα empty shell, όπως είπατε κι εσείς Θέλουμε λοιπόν να, να αναπτύξουμε κάποιες ιδέες κάποιες συστάσεις για τις αρχές για να μπορέσουν να τι εφαρμόσουν. τη βασική ιδέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει το counterparty risk management. Ε, αυτό γίνεται εκεί όπου βρίσκεται βεβαίως ο πελάτης. Ο κίνδυνος για την αγορά μπορεί να έχει να κάνει με τη μητρική εταιρεία, με τη μητρική οργάνωση, αλλά η εποπτική αρχή εντός της Ευρώπης 27 πρέπει να έχει πρόσβαση ε, στις κατάλληλες πληροφορίες για να μπορέσει να αξιολογήσει ε, την, την διαχείριση του κινδύνου και το πόσο, κατά πόσο αυτή λαμβάνει η χώρα καταλήλως. Επίσης εξετάζουμε τη δυνατότητα ενός σοκ. Ε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιους κινδύνους τοπικά όταν συμβεί κάποια ακραία απόφαση, έχουμε ένα σοκ. Υπάρχει λοιπόν θέμα ορατότητας του κινδύνου για την αγορά από τις τοπικές αρχές και να μπορεί εφόσον υπάρξει κάποια κρίση ε, να αντιδράσει έγκαιρα αυτή η αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Δελβό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση προς τον κύριο Μέγιο. για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των ΕΖΑΣ. Αυτά τα οποία είπε μου προκάλεσαν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι υπάρχει συνεπώς μια κάποια συνένεση και μετά από χρόνια εμπειρίας τα οποία έχουμε συλλέξει θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την συνεκτικότητα και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά φυσικά δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Υπάρχει μια κάποια νευρικότητα σε σχέση με τις ε, διαδικασίες αδειοδότησης ε, ρυθμίσεων μέσω εξουσιοδοτήσεων. Οι επιχειρήσεις υπογραμμίζουν ότι οι προτάσεις αυτές δημιουργούν γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις όταν ένα ταμείο τέτοιο επενδυτικό θέλει να εξάγησε εισαγωγικά τις δραστηριότητες του σε τρίτες χώρες, τα επίπεδα γραφειοκρατίας είναι ιδιαίτερα έντονα. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι ότι αυτού του είδους η παρατήρηση ανήκει στη συνηθισμένη γκρίνια των αγορών ή είναι κάτι το οποίο ενέχει στοιχεία αλήθειας. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο θέμα, λέει η κυρία Ντελβό. Πράγματι εκφράζονται πολλές ανησυχίες από τους διαχειριστές κεφαλαίων για την γνωμοδότησή μας για τις εξουσιοδοτήσεις. Ο λόγος για τον οποίο εκδώσαμε τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση είναι ότι μετά από αυτά τα οποία είδαμε και ανταποκρινόμενοι στην αναχώρηση ή αποχώρηση μάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, Προσπαθούν οι Βρετανοί να δουν πώς μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στο εσωτερικό της Ευρώπης των 27. Αυτή η αναζήτηση για ένα νέο χρηματοπιστωτικό κέντρο θα πρέπει να γίνει ε, σε μια κατάλληλη βάση. Υπήρξαν κάποιες κατευθύνσεις από πλευράς ορισμένων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα για το αν είχαν σαν στόχο την σταθερότητα του χρηματοπιστητικού συστήματος ή από την άλλη την προσέλκυση ε, των, ε, των επιχειρήσεων που έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα κέλυφος πλαισίου προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανταφήσουμε όλα να ρυθμίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τελικά κάθε εθνική ρυθμιστική αρχή αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι μια καλή δουλειά στον τομέα και τον διακανονιστικό ε, και της εποπτείας και ακριβώς επειδή έχουμε κατανείμει την εποπτεία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος ο οποίος να ελέγχει κατά πόσον οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τους και εφαρμόζουν σωστά τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Ευρώπη έχει ένα μοναδικό μοντέλο στον κόσμο σε κάποιους τομείς εποπτείας Έχουμε ένα θα έλεγα βασικό επίπεδο προστασίας, αλλά είναι σαφές ότι απαιτείται ένας μηχανισμός έτσι ώστε η ευρωπαϊκή προοπτική να λαμβάνεται υπόψη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους επιπλέον κινδύνους που μπορεί να δημιουργούν ορισμένες αρχιτεκτονικές και σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο καταναλωτών. Το θέμα λοιπόν είναι να έχουμε τρία άτομα γιατί αυτό είναι, δεν ζητάμε κάτι το υπερβολικό. Να υπάρχουν τρία άτομα τα οποία να έχουν έδρα να εργάζονται εκεί όπου έχει έδρα το συγκεκριμένο ταμείο. Αυτό ζητάμε. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το υπερβολικό. Είναι μια προϋπόθεση, είναι μια δικλίδα ασφαλείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και σε εθνικό εποπτικό επίπεδο. Μπάλτς. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη άκουσα, έχουν τεθεί κάποιες από τις ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω στον Μέγιο αλλά να επανέλθω στην τελευταία ερώτηση της κυρίας Ντελβό και σε σχέση με το Brexit. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς εσείς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΣΜΑ ενώ ε, το Brexit ε, βρίσκεται πρώτων θυρών. Νομίζω λοιπόν ότι Ίσως και οι δύο συμπρόεδροι σας θα μπορούσαν να μας δώσουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και της ΕΣΜΑ για το συγκεκριμένο θέμα. E Αναφερθήκατε στο CCP, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ με τη σειρά μου στον έλεγχο των CCP Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει συζητηθεί. Νομίζω ότι ίσως εδώ να υπάρχει και σύγκρουση αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΣΜΑ και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή προσπαθεί να κάνει κάποιες προτάσεις οι οποίες όμως δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και θα ήθελα να μάθω πώς εσείς βλέπετε τα πράγματα. On Σχετικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα για το Brexit και σχετικά με την αναθεώρηση της ΕΣΑ, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία και το είπαμε πριν από το Brexit, ότι ο μηχανισμός τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι ο πλέον κατάλληλος έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να ρυθμίσει την αλληλοεπίδραση που έχει με τις ομόλογες αρχές. Όταν βλέπουμε εμείς προέρχονται, βλέπουμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που προέρχονται από μια τρίτη χώρα, θα πρέπει να είμαστε σε θέση, σε εποπτικό επίπεδο να δώσουμε μια απάντηση. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς φυσικά με τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές σε όλο τον κόσμο αλλά από την άλλη δεν υπάρχουν οι ίδιες προτεραιότητες κινδύνου στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Πρέπει εδώ να υπάρξει μια μορφή ελέγχου των αντιστοιχειών θα έλεγα και το πρόβλημα αυτό ε, χειροτερεύει με το Brexit γιατί βλέπουμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό χρηματοπιστωτικό κέντρο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πάντα πολύ σημαντικό για τις 27 χώρες. Συνεπώς λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα ρυθμιστεί και από, τους, από τις εποπτικές αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το θέμα δεν είναι οι επικαλύψεις, το θέμα δεν είναι οι ατέλειες, το θέμα είναι να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε εγκαίρως τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργούνται για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι από τους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνει η έκθεση της ΕΣΜΑ. και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή πριν ε, φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο έτσι ώστε ο μηχανισμός να είναι σε θέση να λειτουργήσει πριν ολοκληρωθεί ε, το Brexit. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Όπως και ο Αντρέα έλεγε προηγουμένως, είπε ότι μπορεί να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων θα μπορούσε να ισχύσει και για μένα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η αδίποτε λύση μπορούμε να βρούμε, η λύση αυτή θα πρέπει να είναι λειτουργική, να υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες στις αγορές να γνωρίζουν πραγματικά την ιεραρχία στις αγορές, ποιοι είναι υπεύθυνοι και γιατί. Είναι πάρα πολύ περίπλοκη η διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε εκτελεστικό επίπεδο και σε σχέση με τη νέα εκτελεστική επιτροπή. Σε πάρα πολλές αποφάσεις απαιτείται ε, να ε, υπάρχει συμφωνία και γνώμη και της Κεντρικής Τράπεζας Εκδόσεων και της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν οι συμμετέχοντες στις αγορές, οι καταναλωτές να γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνο και γιατί. Να πω επίσης ότι ένα μεγάλο κομμάτι των παραγόγων ε, δεν είναι αποκλειστικά μόνο ε, για, ε, τις, για ομόλογα. Εγώ καταλαβαίνω το θέμα της Κεντρικής Τράπεζας Εκδότριας. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο ΦΕΤ και στο CSTC και εμείς δείξαμε σαν έσμα, έχω την εντύπωση, ότι έχουμε δουλέψει καλά και σε σχέση με το ΕΜΙΡ. Έχουμε ξεκινήσει επίσης και τα πρώτα stress test για τις e CCP και νομίζω ότι η εμπορογνωμοσύνη αυτή μπορεί να ληφθεί πλέον υπόψη. Ε, φυσικά η εποπτεία από τη μία και ο διακανονισμός και οι ρυθμίσεις από την άλλη είναι δύο διαφορετικά πράγματα, προσθέτει ο κύριος Γκουαλτιέρη. Είναι βασική αρχή της δημοκρατίας. Η κυρία Μπερές. Όχι, δεν θέλει κύριε Μπερές. Είναι αγγίλ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, οι πτήσεις καθυστέρησαν. Αλλά θα ήθελα να τονίσω αυτό το οποίο μόλις άκουσα. Τις πρόσφατες προτάσεις και την αναθεώρησή τους και βεβαίως την εποπτεία των τρίτων χωρών. Υπάρχει λοιπόν σαφής αύξηση στον υποπτικό ρόλο της ΕΣΜΑ και υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους η ΕΣΜΑ έχει νέες αρμοδιότητες και υπάρχουν και ερωτήσεις για τους πόρους και την ικανότητα να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Το θέμα ήταν ότι αντιλαμβάνομαι την ε, ανησυχία σας ε, για... Ποιος το λένε τώρα. Τους επόπτες ε, τρίτων χωρών. Αλλά... Και το ότι θέλετε και άλλους πόρους, αλλά τι άποψη έχετε για την πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά την πολιτική την εδαφική της ε, Κομισιόν. Ε, αυτό σημαίνει έχει κόστος για εσάς και για τους άλλους. Ε, θεωρείτε ότι έχει σημασία να διατηρηθεί αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα το οποίο αφορά όλες τις εποπτικές αρχές. Για υπό μίαν έννοια το Brexit θα διευκολύνει μια πιο ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή εποπτεία. δεν ξέρω εάν μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά εσείς ως ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Και τέλος να αναφερθώ στον κύριο Ένρια της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Τραπεζών. Βεβαίω. η βιώσιμη χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό θυμό, όμως η ομάδα υψηλού επίπεδου της ε, Κομισιόν κατέληξε ότι πρέπει να δοθούν επιδοτήσεις για την πράσινη χρηματοδότηση. είστε υπέρ, ε, συμφωνείτε με τις ιδέες ε, που ακούστηκαν και από την Ολίβια Γκέρσον που είπε στις 25 Σεπτεμβρίου ότι πρέπει να υπάρξουν κάποια αντικίνητρα για να τιμωρούμε τις επενδύσεις σε ορυκτά κάψιμα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ναι, για το θέμα του να γίνει ένα μεγάλο βήμα άμεσης εποπτείας, εάν μπορούμε να το κάνουμε, τι πόρους χρειαζόμαστε. Νομίζω σε γενικές γραμμές η στελέχωση και οι ενδείξεις που υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε κατελάχιστον, αλλά είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τους πόρους. Νομίζω γενικότερα για το εάν εμείς σαν οργανισμός θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα ήθελα να επανέλθω εκεί όπου ξεκινήσαμε το 2011. Νομίζω τότε υπήρχαν ανάλογες ανησυχίες για το εάν η ΕΣΜΑ μπορεί να δημιουργήσει κάποιους οργανισμούς αξιολόγησης. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν τεράστιες ε, διαφορές ε, μεταξύ των και των δε, αλλά από την άλλη δείχνει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και βεβαίω δείχνει ότι μπορούν να γίνουν αυτές οι αλλαγές των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Για το πού θα βρίσκονται τώρα τα θεσμικά όργανα, όπως ξέρετε η ΕΣΜΑ στο παρελθόν έχει εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να στηρίξει τις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές Εργαζόμαστε ακριβώς το θέμα της ισοδυναμίας για να λειτουργήσουν αυτές οι αγορές και νομίζω πως η ισχύ της πρότασης είναι να, να έχουμε και τις δύο προτάσεις επιτάπητος. Υπάρχει ακριβώς η δυνατότητα ισοδυναμίας και επιπλέον έχουμε και αυτές τις αυξημένες εποπτικές αρμοδιότητες και ακριβώς ε, δικαίως έχουμε και τις δύο επιλογές ανοιχτές γιατί δεν ξέρουμε πώς θα πάει η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασιλείο. Παραδείγματος χάρη. Ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να είναι σαφές είναι η πρόσβαση στις εποπτευόμενες ε, οντότητες εκτός της Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει κάποια αξιοπιστία, πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε σε κάποιο μοντέλο όπου ε, έχουμε κάποια υποδομή εκτός της Ένωσης, η οποία θα είναι πολύ σημαντική για την Ένωση. Ευχαριστώ, Βέρνερ Λάγκεν. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να μας δοθεί ένας ρόλος ε, στον τομέα της ε, βιώσιμης χρηματοδότησης, τον οποίο τώρα δεν έχουμε μέχρι στιγμή. Σε γενικές γραμμές νομίζω βεβαίω ε, θα το στήριζα. Καλό είναι να μπούμε σε αυτόν τον τομέα. Σε γενικές γραμμές είμαι κάπως επιφυλακτικός όταν μιλάμε για την αλλαγή της αξιολόγησης κινδύνου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να στηριχθεί ένας κλάθος. Πρέπει να είμαστε ουδέτεροι ως προς τον κίνδυνο. Ε, εκεί πέρα είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στο μέλλον. Κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια γενική ερώτηση προς τρεις πρόεδρους. Τα συγκεκριμένα παραδείγματα από το θέμα της ΕΙΟΠΑ. Έχω εμπειρία πολλών ετών. Είναι ότι σας τίνουν να ασχοληθούν με θέματα που πηγαίνουν πέρα από το επίπεδο 1 και 2 και έτσι να αποκτήσουν ε, στην πράξη κάποια αρμοδιότητα παρά το ότι δεν απασχολεί ε, κάτι τέτοιο το Κοινοβούλιο. Οπότε έχουμε αυτό το δημοκρατικό κενό το οποίο πρέπει ε, να γεμίσει. Αυτό το δημοκρατικό κενό κατά την άποψή μου πρέπει να παραμείνει όσο δυνατόν μικρότερο το έλλειμμα αυτό εάν θέλετε. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο όταν το ζητάνε δύο τρίτα των ενδιαφερομένων. Αλλά αυτό δεν επαρκεί κατά την άποψή μου. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι μηχανισμοί ελέγχου για δραστηριότητες επίπεδου 3 είναι ανεπαρκείς και πρέπει να βελτιωθούν. Θα δώσω παραδείγματα από τον τομέα του κυρίου Μπερναρντίνο ή ΑΙΟΠΑ. Παρά το ότι ο συνομοθέτης δεν έχει εγκρίνει ακόμα τα μέτρα επίπεδου 2, π.χ. στο IDD, η ΑΙΟΜΠΑ ανέλαβε πρωτοβουλία που ε, ρητός ε, και συνειδητά δεν περιέλαβαν οι συνομοθέτες και ήδη στο παρελθόν η ΑΙΟΠΑ πάντα έθετε ζητήματα επίπεδου 3, π.χ. το τελευταίο ζητήματα για το πώς θα έπρεπε να υποπτεύεται μία ασφαλιστική εταιρεία. Και κύριε Βερναντίνο, ίσως το γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι είχατε αναπτύξει με ίδια πρωτοβουλία 7.000 σελίδες ε, για αρμοδιότητες ε, σχετικές. Λοιπόν, και προς τους τρεις ε, απευθύνομαι. Πώς κρίνετε τις δυνατότητες ελέγχου για μέτρα επίπεδου 3. Και ο κύριος Μπερναρντίνο. Ευχαριστώ και εγώ και τον κύριο Λάγκεν για την ερώτησή του. και το θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών και το θέμα των ρυθμίσεων τρίτου επίπεδου είναι κάτι το οποίο μας απασχόλησε. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις, ε, uh, τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες και την οδηγία που τις διέπει οι κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες προτείνουμε εμείς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα συμβατές με αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις οδηγίες μέχρι τώρα. Και όπως είπα στην παρέμβασή μου, είμαστε απογοητευμένοι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έλαβε πλήρως υπόψη αυτά τα οποία είχαμε εμείς προτείνει. Ε, οι επιχειρήσεις οφείλουν να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και να είναι διαφανείς στη διαχείριση των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων έτσι ώστε να προωθηθεί το συμφέρον των καταναλωτών. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για τις ελεγκτικές διαδικασίες που προβλέπονται στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ανήκει και στα δικά μας επίπεδα ελέγχου. Εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συζητήσουμε μαζί σας με διαφορετικούς τρόπους και κάτω από διαφορετικές καταστάσεις το τι πραγματικά κάνουμε. Είμαι πεπισμένος ότι οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα απόσπαστο στοιχείο εξασφάλισης της συνοχής των στοιχείων που συλλέγουμε. και νομίζω ότι δεν είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργούν το πρόβλημα. Αν δεν υπήρχαν οι κατευθυντήριες γραμμές θα υπήρχε ένα patchwork εθνικών ρυθμίσεων εφαρμόσιμων ταυτόχρονα στις ίδιες περιπτώσεις. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ κακό για την εσωτερική αγορά. Σχετικά με τις ελεγκτικές διαδικασίες όπως προβλέπονται από τις κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί θα πρέπει φυσικά να διατηρούμε πάντα την πλήρη ελευθερία μας, αλλά δεχόμαστε προτάσεις οι οποίες να δίδουν στο συνολικό πλαίσιο μια καλή ισορροπία. Νομίζω ότι και οι ομάδες ενδιαφερόντων θα μπορούσαν να θέσουν κάποια θέματα ε, εάν θεωρούν ότι εμείς ξεπερνούμε την εντολή την οποία έχουμε αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για μια σωστή σύνθεση των ομάδων συμφερόντων. Νομίζω ότι είναι περισσότερο κλείνει προς τις ε, επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή η ισορροπία και γι' αυτό ίσως θα πρέπει να αποκατασταθεί. Επίσης υπάρχει και η Επιτροπή Εφέσεων, το Συμβούλιο μάλλον Εφέσεων, ε, και εκεί μπορεί να ελεγχθεί το εάν πράγματι εμείς ε, σεβόμεθα τις αρμοδιότητές μας και αν μένουμε μέσα στο εσωτερικό του πλαισίου που προβλέπεται για αυτές. Λοιπόν, νομίζουμε ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, είναι καθοριστικές για τη συνοχή των ελεγκτικών και εποπτικών διαδικασιών. Είναι σημαντικά τα θέματα αυτά. Πάντα μπορεί κανείς να έρχεστε σε επαφή μαζί μας, να μας ζητάτε να ερχόμαστε εδώ και να σας εξηγούμε το τι πραγματικά κάνουμε. Δεύτερον, ξεκάθαρα και σκόπιμα, εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας πάντα στα πλαίσια του επίπεδου 1. Είναι η καλύτερη μορφή προστασίας για οποιοδήποτε νομικό κίνδυνο που μπορούσε να δημιουργηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς ε, θα μπορούσα να έχω ένα μετρητή ε, στο γραφείο μου το οποίο να καταγράφει κάθε φορά που λέω στο προσωπικό μου ότι πρέπει να εμείνουν αποκλειστικά στο επίπεδο 1. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθήκων θα πρέπει να ελέγχουν αυτά τα οποία κάνουν οι εποπτικές αρχές, αυτά τα οποία κάνει η ΕΣΜΑ και αν είναι συμβατά με το επίπεδο 1. Τώρα, αν είμαστε σε θέση να είμαστε κοντά στο επίπεδο 1 και να έχουμε και περισσότερα στοιχεία τα οποία να κατανοήσουμε καλύτερα, να μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα, γιατί όχι. Θα ήθελα επίσης ε, να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε διαθέσιμα και τα τρία επίπεδα. Όταν υπάρχουν και τα τρία επίπεδα είναι καθοριστική καθοριστικό στοιχείο της επιτυχίας μας. Και στα πλαίσια των ερωτημάτων που τίθενται πάρα πολύ συχνά, μας ζητούν κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Ένα τομέα στον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργία μα είναι το ποια θέματα αντιμετωπίζονται σε ποιο επίπεδο. Αλλά αυτό είναι μια συλλογική ευθύνη, Το τι ανήκει και γίνεται στο ένα, το τι ανήκει και γίνεται στο δύο και το τι ανήκει και γίνεται στο 3. Αυτό δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι θέλουμε περισσότερες εξουσίες. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις δικές σας νομοθετικές ρυθμίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας δώσω ίσως κάποια παραδείγματα εδώ. Εμείς ξεκινήσαμε με τις κατευθυντήριες γραμμές πρόσφατα για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας και των ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων γενικότερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε κεντρικό επίπεδο και είναι ένα σταθερό αίτημα από πλευράς των εθνικών εποπτικών αρχών. Thank you, Η κυρία Μπερές τελευταία, αλλά ο πόσο σημαντική. Και δεν την ερώτηση από το στόμα κύριε Μαγιόρ για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα CCP. Θα ήθελα να αναφερθώ στην αναθεώρηση του άρθρου 22 του, του καταστατικού του, της ΕΚΤ. Πιστεύετε ότι αυτό οδηγεί σε μια σωστή ισορροπία, ότι αφορά τι εξουσίε που προκύπτουν από τα CCP. Κύριε Εντρία, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του CRR, γίνεται μια συζήτηση στο Συμβούλιο βεβαίω, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα, θα μα έρθει και εδώ στο Κοινοβούλιο για τα άρθρα 7 και 8 της CRR και για τα waiver ή τα liquidity, μας περιπτώσει. Ε, εσείς τι πιστεύετε για τα άρθρα 7 και 8 και για τη δημιουργία μιας ενός κεφαλαίων που να έχει μια υπερεθνική δυνατότητα. Ε, και κύριε Μπερναρντίνο, τέλος μου είπαν ότι υπάρχει μια πρακτική κάποιων ασφαλιστικών εταιριών που είναι εγκαταστημένες αυτή τη στιγμή στο Γιβραλτάρ. Έχετε ασχοληθεί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και σα ευχαριστώ για αυτό. σα είχα ρωτήσει σχετικά για το Γιβραλτάρ όμως οπότε ακούω υπάρχει μια είδου αυτονομία όπου οι άδειε δεν χορηγούνται από το Λονδίνο αλλά το Γιβραλτάρ εν τη σοφία του χορηγεί αυτέ τι άδειε και σε επίπεδο dumping ε, είμαστε αρκετά ψηλά, έτσι. Και τελευταίο ερώτημα για σας, ε, τηλεγραφικά βέβαια όλα αυτά, έτσι δεν έχουμε χρόνο, το ξέρω. Ε, εκθιάζεται πολύ το BEPS. Βεβαίως ε, υπάρχει lobbying έντονο προς εμάς, μην ανησυχείτε. Και το πρώτο επιχείρημα είναι ότι, ξέρετε, πρέπει οπωσδήποτε να επιτρέψουμε την ε, ε, την έξοδο των κεφαλαίων, διότι δεν, ε, οι ραντιέρδες, σε πάση περιπτώσει, ε, είναι πλέον ξεπερασμένο πράγμα. Αλλά μπορεί, μπορούμε να μετατρέψουμε την αποταμίευση των ε, συνταξιούχων σε ένα αμυγός επενδυτικό προϊόν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντελού. Ναι, για τα liquidity waivers, ακούστε, δεν έχουμε επίσημη θέση της CBA, αλλά να σας πω τη δική μου. Είναι σημαντικό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης διαπιστώσαμε ότι πέρθηκαν πολλά μέτρα ε, που οδήγησαν σε κατακαιρματισμό Πρέπει λοιπόν να στείλουμε ένα μήνυμα για μια καλύτερη διασυνοριακή τραπεζική δραστηριότητα την Ένωση. Ε, και βεβαίω η διαχείριση τη ρευστότητα είναι ένα σημείο κλειδί εδώ και Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξία στα κράτη-μέλη ό,τι αφορά τη μεταβίβαση κεφαλαίων και ρευστότητα όταν έχουμε να κάνουμε με κοινέ αποφάσει για τα κεφάλαια και τη ρευστότητα. Είναι σημαντικό αυτό και βεβαίω τα waivers αυτά μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει να ε, βελτιωθεί η ολοκλήρωση τη αστική αγορά είναι επανέλθει η ολοκλήρωση τη αγοράς αγορά. Να, να είμαι σύντομο για τα δύο ερωτήματά σα για τον Γιβραλτάρ πρώτα. Είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε βέβαια. Διότι το Γιβραλτάρ αποτελεί μέρο τη εσωτερική αγορά. Ισχύουν εκεί οι κανόνε περί και υπάρχουν πολλέ εταιρείε βεβαίω που ε, συναλλάσσονται διασυνοριακά έχουμε συνεργαστεί μαζί τους. Κάποιες από τι πλατφόρμες τις οποίες αναφέρθηκα σε ό,τι αφορά τις δυσνοριακές επιχειρήσεις ε, έχουν εμπλακεί σε ιστορίες με τον Γιβραλτάρ. Έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά. Είχαμε σημαντική παρέμβαση ε, με τις εποπτικές αρχές ε, της χώρας υποδοχής και της χώρας προέλευσης. Ε, είμαστε σε στενή συνεργασία με την αρχή του Γιβραλτάρ για να είμαστε βέβαιοι ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο θα εφαρμόζεται πλήρω είναι κεφαλαίωδες αυτό. Ε, έχουμε πραγματικά στους τελευταίους μήνες δαπανίσει πολύ χρόνο να συζητούμε μαζί τους. Τώρα για το ΠΕΠ. Ε, Βεβαίω θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες να το συζητήσουμε το ΠΕΠ με το Κοινοβούλιο για την συσσόρευση και αυτό που αναφέρατε. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Το ΠΕΠ πρέπει να είναι ένα ε, μακροπρόθεσμο προϊόν αποταμίευσης. Δεν πρέπει δηλαδή, να υπάρχει δυνατότητα ε, κάποιος να μπορεί να πάρει τα χρήματα οποιαδήποτε στιγμή. Υπάρχουν λύσεις γι' αυτό και αυτό να αποτελέσει μέσω κατά τη γνώμη μου ε, αυτής της επιλογής, διότι τελικά αυτή είναι η επιλογή που θα επιλέξουν οι περισσότεροι πολίτες. Ε, υπάρχει ένα επιχείρημα εδώ δημόσιας πολιτικής, ε, έτσι ώστε ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου που συσσωρεύεται να πληρώνεται είτε ετησίως ε, ε, και όχι να μπορεί κάποιος άμεσα να το ρευστοποιήσει. Για το ΕΜΙΡ 2,2 και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την παρακολούθηση των CCP είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη βέβαια ε, στο παρόν ε, σύστημα. Οι κεντρικές τράπεζες εκπροσωπούνται δηλαδή στα διάφορα κολέγια αποφάσεων, δείτε και το αμερικανικό μοντέλο. Άλλωστε η Fed έχει ένα πολύ κεντρικό ρόλο. Ταυτόχρονα το άρθρο 22 του καταστατικού ε, δημιουργεί κάποιε ανησυχίε. Αυτό σχετίζεται και με το προηγούμενο θέμα που συζητήσαμε. Πρέπει να ξέρουμε να είναι σαφέ ποιο είναι υπεύθυνο γιατί σε ένα σύστημα. Να μην έχουμε επικαλύψει ό,τι αφορά τι αρμοδιότητε. Και ανησυχώ ιδιαίτερα με το προτινόμενο κείμενο σχετικά με το άρθρο 22. Διότι αναλαμβάνουμε ένα αριθμιστικό ρόλο που είναι παράλληλο με το αριθμιστικό ρόλο τη Κομισιόν, το Συμβούλιο ε, και η ΕΣΜΑ έχει ένα ρόλο στο σύστημα αυτό. Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι ποιε είναι οι ρυθμιστικέ αρμοδιότητε που έχει ο καθένα όταν αλλάζει το ε, καταστατικό σε σχέση και με τι αρμοδιότητε στο ΕΜΙΡ. Ε, πρέπει να είναι σαφέ ε, ποιοι είναι οι συμμετέχοντε στην αγορά και ποιο είναι υπεύθυνο. Κατά τη γνώμη μου δεν θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα αριθμιστικό ανταγωνιστικό ή να έχουμε ανταγωνιστικά αριθμιστικά συστήματα μεταξύ του. Πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση βέβαια ε, αλλά το κείμενο αυτό θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και θα πρέπει να είναι και ε, βιώσιμο, μακροπρόθεσμα. Ακόμα και το να αλλάζουν ε, τα πρόσωπα που παρτίζουν ε, τις διάφορες αρχές. Είναι λοιπόν σημαντικό οποιαδήποτε αλλαγή στο άρθρο 22 να μην ε, συγκρούεται με τις απαιτήσεις ΕΜΗΡ. Επιπλέον Υπάρχει, υπάρχουν και αλλαγές στο ΕΜΙΡ 2,2. Εκεί όπου υπάρχουν απαιτήσει ρυθμιστικές περαιτέρω που προέρχονται από τις κεντρικές τράπεζες, αυτό θα αφορά τρίτες χώρες. Δεν θα αφορά ε, τις χώρες της Ένωσης. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη, πολύ ενδιαφέρουσα η ακρόαση αυτή και βεβαίως θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και θα παραμείνουμε σε επαφή. Διότι έχουμε και νομοθετικές διαδικασίες, ε, ε, αναθεώρηση της ΕΣΑ, τα CCPs κτλ. κτλ. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Κλείνουμε με το σημείο αυτό. Θα δώσω τώρα την Προεδρία στην, στον Αντιπρόεδρο, τον Μάρκους Φέρμπερ. dear colleagues. Uh, ε, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ο χρόνος ε, περνάει, οπότε συνεχίζουμε απευθείας. Ε, περνάμε σε ανακοινώσει του Προέδρου. Ανοιχτή συνεδρίαση συντονισμού. Γεια σας, φίλοι των συντονιστών με τον Κρίστιαν Τίμαν, πρόεδρο της ομάδας ειδικών της αηφόρου χρηματοδότησης, θα γίνει αύριο στις 1.30 ώρα. Σας παρακαλώ να βγείτε ήσυχα από την αίθουσα. Συνεδρίαση θα είναι δημόσια. Λέω τι να πω, ισότα μία κόντων τα λέω. Ανταλλαγή απόψε με εθνικά κοινοβούλια. Υπενθυμίζουμε στους βουλευτές ότι οι εθνικοί βουλευτές θα έρθουν στην ΕΚΟΝ αύριο το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 5.30 πριν από την ψηφοφορία της δεύτερης έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας ε, του εξαμήνου για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, και τη δημοσιονομική στάση των χωρών τους και θα έχουμε άλλη μια ανταλλαγή απόψεων στις 4.30 για μια πρόταση για κοινή φορολογική βάση επιχειρήσεων και ενοποιημένη επίσης. Και βεβαίω δεδομένου του ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια εκφέρουν άποψη από των προτάσεων αυτών, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους εθνικούς βουλευτέ για τις προκλήσεις αυτών των μεταρρυθμίσεων και για την φορολόγηση της ψηφιακή οικονομίας. Μετά έχουμε περίληψη αποφάσεων και συστάσεων των συντονιστών τη 5 η Οκτωβρίου κατανομή εκθέσεων πρώτα απ' όλα για τις τρεις ρυθμιστικές αρχές ε, και τις αλλαγές στους άλλους τομεακούς κανονισμούς που δεν θα αναφέρω. Αυτά πάνε σε ΕΛΚ και Σοσιαλδημοκράτες. Δεύτερον, οδηγία που τροποποιεί την οδηγία ΜΥΦΙΔ και Φερεγκαιότητα 2 πηγαίνουν στο ΕΛΚ και Σοσιαλδημοκράτες και πάλι για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας και πάλι ΕΛΚ και Σοσιαλδημοκράτες από κοινού. Για, συντονι... για δημοσιονομικό συντονισμό 2018 και Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πάει σοσιαλδημοκράτες, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο ΕΛΚ και οποία έκπληξης ή αηφόρος χρηματοδότηση πράσινου. Γνωμοδοτήσει, ανταγωνισμό ε, ανταγωνισμός αερομεταφορές φιλελεύθερους, ε, στο Προεδρείο πηγαίνουν τα τέλη βαρέων οχημάτων, ε, απαλλαγή της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής στο Προεδρείο, απαλλαγή της ΕΙΟΠΑ επίσης, απαλλαγή της ΕΣΜΑ επίσης στο Προεδρείο και πλαίσιο για τον έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει στο ECR. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο του χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων. Θα σας ενημερώσουμε τους συντονιστέ για το τι θα γίνει και αυτοί θα ενημερώσουν τους συνάδελφου οι συντονιστές συμφώνησαν να ζητήσουν άδεια για κάποιες έκτακτες συνεδριάσεις πριν από το τέλος του έτους, συγκεκριμένα 5η 23 Νοεμβρίου το πρωί, Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου αργά το απόγευμα, βράδυ βασικά από τις 7 μέχρι τις 8.30. Α, όχι, δεν είναι 4 Δεκεμβρίου Στρασβούργο και 5η 3 Δεκεμβρίου το πρωί αποστολές του 2018 αποφασίσαμε να γίνουν οι εξή αντιπροσωπείες το 2018. Πρώτα απ' όλα επισκέψεις ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πρώτο εξάμεινο, δεύτερο εξάμεινο στην, στη δεύτερο τρίμηνο, με στην ε, Βασιλεία και στην Διεθνή Ένωση Υποπτικών Αρχών Ασφαλιών, Γαλλία. Επίσης ε, το πρώτο εξάμεινο, Ιταλία δεύτερο εξάμεινο, Ουάσιγκτον 5 με 20 Ιουλίου, Κίνα 17 με 21 Σεπτεμβρίου, Ελπίζουμε του χρόνου να τα καταφέρουμε, γιατί είχαμε ήδη οργανώσει κάτι και ετήσια συνεδρίαση του Δελτανιτάφου που λάβει χώρα, που δεν θα είναι στην Ουάσιγκτον, από 10-14 Οκτωβρίου στο Μπαλί για όσους δεν γνωρίζουν. Όσον αφορά τις αποστολές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι συντονιστές συμφώνησαν να στήσουν μία ή δύο έξτρα θέσεις ανά αποστολή ακροάση 2018 συμφωνήσαμε να υποβάλουμε τον εξής κατάλογο στην διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών. Το μέλλον της ε, ΟΝΕ, μεταρρύθμιση ΕΖΕ και Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας, ΕΜΙΡ και Κανονισμός Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, παραπλανητική διαφήμιση χρηματοπιστωτικών προϊόντων και φορολογία, ορισμός μελών του ΔΣ του ESGB ε, θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Επιτροπής και επίσης να βρεθεί η κατάλληλη ημερομηνία για ακροάσεις υποψηφίων. Σημείο 6. Δύο οργανικές διαπραγματεύσεις. Ε, ο πρώτος τριμερής διάλογος στις ε, 3 Οκτωβρίου. Όχι, ο 7ος ΝΑΤΟΣ, ναι. Ο έβδομος διάλογος για την πέμπτη οδηγία ε, έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τα, συζητήθηκαν τα εξή ε, πραγματικοί ιδιοκτήτες και πληροφορίες περί αυτών, πολιτικά πρόσωπα, χρυσές βίζες και διαβατήρια, κριτήρια για ε, τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, άρθρα 6, 63 και 54 έλεγχοι αρμοδιότητες αρχών χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και συνεργασία αυτών η ημερομηνία μεταφορά στην νομοθεσία και μεταβατικές περίοδοι. Επίσης, οι Επίτροποι συζήτησαν ένα νέο πακέτο προτείνει η Εστονική Προεδρία οι συνομοθέτες διαπίστωσαν ότι έγινε, σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος. Ο επόμενος τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 14 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Για την οδηγία κεφαλιακής επάρκεια και τις μεταβατικές διατάξεις 28 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου έλαβαν χώρα και για τα IFRS 9. Καταλήξαμε σε συμφωνία για τις μεταβατικές διατάξεις για τη μεγάλη έκθεση, όμως δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος για τα πρότυπα IFRS 9. Οι συνομοθέτες είχαν ριζικά διαφορετικές απόψεις για το ποια προσέγγιση έπρεπε να ακολουθηθεί για να υπολογιστεί το ποσό το οποίο θα έπρεπε να προσθεθεί και απορρίφθηκε από το Συμβουλίο Συμβαστική Πρόταση του Κοινοβουλίου. Η επόμενη συνεδρία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου. Ερχόμαστε στο σημείο 7. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δίνω τον λόγο στον Λούντεκ Μάιερ, τον οποίο αντικαστά Μπορκάρτ Μπάλτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητά συγγνώμη ο Λούντιχ για την αποψία του σήμερα και μου ζήτησε να παρουσιάσω την πρόταση αυτή εξ ονόματός του επί τη βάση των ερευνών που έκανε ο Λούντε και μετά από την ενδιαφέρουσα επίσκεψη που έκανε στην έδρα της τράπεζας στο Λουξεμβούργο θέλει να υπογραμμίσει τη σημασία της Τράπεζας Επενδύσεων για την απακατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία σε επίπεδα προκρίσης. Είναι απαραίτητο όμως να ανακατευθύνουμε σωστά τις δραστηριότητες της τράπεζας αυτής για να διασφαλίσουμε την προσθετικότητα όχι μόνο αντικυκλικός ρόλος αλλά και τομείς όπως αποτυχίες των αγορών και άλλοι τομείς που έχουν ε, υψηλό κόστος και ο Λούντεκ θέλει να υπενθυμίσει και τον επίγοντα χαρακτήρα της διευκρίνησης των συνεπειών του Brexit στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. που θα επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της και ο εισηγητής ζητά επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει και να καταγράφει πολύ προσεπτικά τις εντολές και την εκπλήρωση των εντολών τις οποίες έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον τομέα του διοικητικού κόστους. Αυτά όλα χαρακτηρίζουν και την ανταγωνιστικότητά της. Και τέλος ο Λούντεκ θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει, να δοθεί προτεραιότητα στις εξωτερικές δράσεις σε τομείς υψηλής ε, σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει τεράστια δυνατότητα για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας να βελτιώσει την κατάσταση στην Ουκρανία η οποία χαρακτηρίζεται από αστάθεια λόγω ακριβώς ε, της σύγκρουσης ε, με την συμμετοχή δυστυχώς και των στρατιωτικών υπηρεσιών της Ρωσίας. Είναι δεκτικός στις παρατηρήσεις σας και στις τροπολογίες σας, οι οποίες αναμένει βεβαίως ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκθεσής του. Ευχαριστώ κύριε Μπάλτς. Περνάμε στους σκιώδης ο Χαουρέγγι για τους ε, σοσιαλιστές. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγήτη τον κύριο Νίτερ Μάγερ. Σε γενικές γραμμές η έκθεσή του είναι μια καλή βάση για να έχουμε μια καλή συνεισφορά ως Επιτροπή Εκόν Τρία σχόλια έχω να κάνω. Θα τις αναφέρω στο όνομα της ομάδας μου μέσω των τροπολογιών βέβαια. Πρώτον, σε σχέση με τη φιλοσοφία που μόλις εκφράστηκε για τον, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον οικονομικό κύκλο ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η επιρροή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να επανέλθει η, η ανάπτυξη δεν ε, καλύπτονται στα σημεία 3 και 4 της έκθεσης Εκεί λέμε ότι η αντικυκλική αυτή η λειτουργία έχει τελειώσει. Εμείς δεν είμαστε υπέρ ε, του να λέμε κάτι τόσο ε, έτσι απόλυτο. Διότι ο προπολογισμό παραμένει αρκετά αδύναμος. Ο Η δημοσιονομική κατάσταση είναι ε, Δεν υπάρχει επίσης προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Και το χάσμα στις επενδύσεις ε, πριν από την κρίση και μετά την κρίση δεν έχει κλείσει. Εξακολουθούν να υπάρχουν λόγοι λοιπόν ε, να είναι, να είναι φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με, να είναι αποτελεσματική αλλά να δρά. Στο σημείο 8 μάλιστα γίνεται αναφορά στην ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ό,τι φορά την εφαρμογή του σχεδίου Juncker. Ε, και αυτό είναι ακριβώς που δίνει αυτήν την απέτηση η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, να παραμείνει στην πρώτη γραμμή. Γιατί χρειάζεται, χρειάζεται για τι επενδύσει. Το δεύτερο που θέλω να πω έχει να κάνει με το Brexit. Ο εισηγητή αναφέρθηκε στην ανάγκη να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις του Brexit στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, θα πρέπει εμεί να είμαστε κάπω πιο συγκεκριμένοι όμω σε ό,τι αφορά το πώ σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τι επιπτώσει του Brexit για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει η Επιτροπή ΕΚΟΝ ενδεχομένω να αναφερθεί στην δυνατότητα να αγοράσουν οι λοιπές χώρες ε, τις μετοχές, εν πάση το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου, για να μην χαθούν χρήματα κάτι παραπάνω πρέπει να πούμε, δηλαδή, πέρα από δύο γραμμές που λέμε για τον Brexit. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε ποιο θα είναι το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε ε, μετά τον Brexit, με το βρετανικό κεφάλαιο. Στην παράγραφο 7 τώρα γίνεται μια αναφορά στην σημασία των εξωτερικών επιχειρήσεων και εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Πιστεύω ότι η ΕΤΕ έχει ένα ρόλο να παίξει όχι μόνο στην Ανατολή, γιατί αναφέρθηκε η Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στη Μεσόγειο, στην Αφρική. Ε, είναι πολύ σημαντικές τις περιοχές ε, από γεωπολιτικής πλευράς για μας και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια αναφορά εδώ ε, στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε αυτήν την Ήπειρο. Και η Λατινική Αμερική βεβαίως είναι πολύ σημαντική. Η παρουσία της ΕΤΕ εκεί είναι σημαντική και λειτουργεί και πολύ, και πολύ καλά οι σχετικές επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναφορά σίγουρα στη Μεσόγειο και στην Αφρική πάντως. Αυτά θα υποβάλουμε τι τροπολογίες μας και θα συζητήσουμε με τον εισηγητή για να έχουμε τελικά μια έκθεση όσο γίνεται πιο συνενετική. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για το ECR δεν είναι εδώ ο κύριος Φόξ. Για τους ε, φιλελεύθερους, Πίτερ, όχι ο Τρεμόζανς και ο εισηγητής, Εντάξει, πράσινη τότε. Μόλις Κορκέιτ. Ναι, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι από το ECR σήμερα να συζητήσουμε για τις επιπτώσεις του Brexit στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος πάντων, ούτε για το ψήφισμα ήταν εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Τι να, πω, τι να πει κανεί. Ε, τέλος πάντων, εγώ παραμένω ε, μια Ευρωπαία πολιτικός, δεν με έχει ακόμα καταπιεί το Brexit. Ε, είναι πολύ σημαντική ε, σημαντικό θεσμό η ΕΤΕ, διότι ε, παρέχει επενδύσει για τη βελτίωση των κοινωνιών μα. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε την ΕΤΕ να επενδύσει στους τομεί εκείνους ε, που θα είναι υποφελεί για του Ευρωπαίου πολίτε. Συμφωνούμε ήδη νωρί στην διαδικασία με πολλά από τα στοιχεία τη έκθεση του εισηγητή. Επίση, η έκθεση αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να παίξει, μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο εκεί όπου έχει αποτύχει η αγορά όταν επενδύουμε σε project με συγκεκριμένα ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, τα οποία δεν είναι ε, όμως ε, ελκυστικά για τους ιδιωτικούς φορείς, μπορεί η ΕΤΕ να καλύψει ένα κενό που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια λόγω υποχρηματοδότησης από τα δημόσια ταμεία. Θα πρέπει βεβαίως η ΕΤΕ να αναλάβει κάποια ρίσκα για να το κάνει αυτό. Θεωρούμε ότι η έκθεση μπορεί να ενισχυθεί σε μια σειρά από και θα πρέπει να δοθεί έμφαση Ιδιαίτερα, παραδείγματο χάρη, στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζήτηση επενδύσεων ε, από μόνη τη. Τα κράτη-μέλη μόνο μπορούν να το κάνουν αυτό. Ατομικά και συλλογικά, λαμβάνοντα αναλαμβάνοντας ε, ε, μάλλον πρωτοβουλίες σε δημοσιονομικό επίπεδο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια πιο βιώσιμη οικονομία. Επίσης δεν συμφωνούμε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι προπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι. Όπως είδαμε, οι ε, ε, δημοσιονομικοί δημοσιονομικές προσαρμογές έχουν οδηγήσει σε απώλεια εισοδήματος, σε μείωση μισθών και σε πολλές περιπτώσεις ε, ο, ο στόχος της μείωσης του χρέους δεν επιτυχάνεται. Χρειάζεται λοιπόν κάποια φορολογικά κίνητρα για να μπορεί να υπάρξει μια όθηση οικονομική για την ανάπτυξη. Τέλος η ΕΤΕ δεν τα έχει πάει τόσο καλά σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Πέτυχε τους στόχους του 25% βεβαίως, αλλά αυτό δεν είναι αρχικά τη γνώμη μας. Στα 16 κράτη-μέλη της Ένωσης η, ΕΤΕ, η υποστήριξη της ΕΤΕ δεν έφτασε καν στο ελάχιστο του 20%. Οι επενδύσεις για την κλιματική δράση ε, αφορά κυρίως τις πιο ισχυρές οικονομίες και τελικά αυτός είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση 70% της ε, υποστήριξης του ΕΦΣΙ για τους ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχεδόν σε μία χώρα, στο Βέλγιο. Ενώ ένα μεγάλο ποσοστό πάει στη Γαλλία, στη Γερμανία και στη Φιλανδία. Λοιπόν, είμαστε ε, ευχαριστημένοι με το πώς προχωράει η έκθεση αυτή τη στιγμή και βεβαίως θα εργαστούμε με την τροπολογιών με τον Λούντο και την ομάδα του. Ευχαριστώ πολύ για την EFTD τώρα. Ο Μάρκο Βάλι ούτε αυτός είναι εδώ και για την ΕΝΕΦ e η Μπάρμπαρα Κάπε αλλά βλέπω ο, είναι Γκίλα έχει στήσει το λόγο η Νίνα Γκίλα μάλλον για το Brexit θα μας πείτε Μακάρι να μπορούσα να σας διαφωτίσω για το Brexit δεν μπορώ όμως για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όμως έχει σημασία το Brexit και δεδομένου του μεριδίου του Ηνωμένου Βασιλείου στην τράπεζα χρειάζεται νομική βεβαιότητα για τα τρέχοντα έργα που χρηματοδοτεί η τράπεζα. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν πολλά έργα και στην ε, περιφέρεια μου που είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να δούμε για να δούμε και ποια είναι η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον ε, προϋπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε στην έκθεση αυτή πως οι εξωτερικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται να, εξωτερικές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά όχι μόνο αυτές, όχι μόνο το τι χρηματοδοτεί στην Ουκρανία. Πρέπει να δούμε την επέκταση της εντολής εξωτερικού δανεισμού, το οποίο έχω καλύψει στην άλλη επιτροπή που συμμετέχω, την Επιτροπή Εξωτερικών που προτείνει η Κομισιόν. Ένα σημαντικό βήμα δηλαδή για να ενισχυθούν οι δραστηριότητες στην νότια γειτονία όπως ε, και το σχέδιο του, της αντιμετώπισης των αίτιων ε, της μετανάστευσης. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε όχι μόνο τις προενταξιακές χώρες ε, και την νότια γειτονιά, και την Μεσόγειο αλλά και την Λατινική Αμερική όπως ήδη αναφέρθηκε και την Ασία. Νομίζω λοιπόν πως ένας βασικός επενδυτής ε, στα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ηγείται δια του παραδείγματος ή την Τράπεζα Επενδύσεων και να μην κάνει επιχειρήσεις και έργα σε φορολογικούς παραδείσους και να εστιάζει πολύ περισσότερο στην βιώσιμη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Ολιβιέντε Μπαντ ε, επικεφαλής ε, της ε, σχετικής μονάδας στο Γραφείο Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σύντομα, σας παρακαλώ. Many thanks, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας δώσατε τον λόγο και ευχαριστώ και τους συγητές και σκιώδεις συγητές για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων να πω σύντομα λίγα λόγια. Πρώτα απ' όλα βεβαίως ε, συμφωνούμε για αυτά τα οποία ακούστηκαν για τον ρόλο της ε, τράπεζας και συμφωνούμε να ενισχυθεί η αξιολόγηση του αντικτύπου. Η προσθετικότητα επίσης είναι πολύ σημαντική διάσταση των δραστηριοτήτων ε, και ακριβώς αφορά την επιλογή έργων και τον τρόπο παρέμβασής μας. Επ' αυτού Προσφάτως ε, αξιολογήσαμε και τον μακροοικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας ε, και του λεγόμενου σχεδίου Juncker και δείχνουμε ότι μέσω του επενδυτικού σχεδίου και των, ε, της κανονικής δραστηριότητάς μας έχουμε σημαντικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Να σας πω κάτι σύντομα, το σχέδιο επενδύσεων και το τι γίνεται για την αξιολόγηση του μακροοικονομικού αντικτύπου το 2020 θα δείτε ότι είχαμε 0,5% και τη δημιουργία 700.000 θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα έλεγα σημαντικός αντίκτυπος. Όσον αφορά τα άλλα τα οποία αναφέρθηκαν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει ενώπιση του νέου πι δελτα και να αναπτύξουμε περαιτέρω το μέσο αυτό και να υπάρχει ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει την χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο μέλλον. Όσον αφορά την διευκόλυνση της εφαρμογής στο επίπεδο των κρατών μελών και του σχεδίου Γιούνκερ αλλά και ευρύτερα για να υπάρχει μια καλή γεωγραφική ισορροπία θα είναι σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις Εθνικές ε, Τράπεζες Ανάπτυξης που βασίζονται στην γνώση της τοπικής αγοράς για να βελτιωθεί ακριβώς ε, η επαφή που έχουμε και βέβαια προσφέρουμε τεχνική αρρωγή για να υπάρξει η προετοιμασία και εφαρμογή των έργων. Θα σταματήσω εδώ για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις σύμβουλές σας. Θα λάβει υπόψη, είμαι βέβαιος, ο εισήγητης αυτά τα οποία είπατε. Προθεσμία η 12η Οκτωβρίου. Η εξέταση των τροπολογιών 6 Νοεμβρίου ψηφοφορίες 20 και 21 Νοεμβρίου και ελπίζουμε να φτάσουμε στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο του 18. Περνάμε στο 8 τώρα. έτσι ώστε οι αρχές του ανταγωνισμού να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά διασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ο κύριος Φάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να το πω καλύτερα από ό,τι τα είπατε εσείς. Πρόκειται πράγματι για ενίσχυση των αρχών ανταγωνισμού και οι συνάδελφοι που είναι εδώ παρόντες, ε, οι σκιώδεις ηγητές δηλαδή βασικά, ε, πραγματικά έχουν την ευγνωμοσύνη μου. Ξέρω πως υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που κολλείονται, έχουν ραντεβού στις χώρες τους κτλ. Γι' αυτό θα περιοριστώ στα ουσιώδη κύριε Πρόεδρε και ελπίζω μετά και εσείς να τα μεταφέρετε στους συναδέλφους που απουσιάζουν <coughs> σήμερα. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω τους στόχους της πρότασης της ε, Κομισιόν. Είναι σωστό ακριβώς οι εθνικές αρχές να ενισχυθούν ε, για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως το δίκαιο του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξυπηρετεί όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ακριβώς ε, θεωρούμε ως Γερμανοί ότι έχουμε μάθει από το παρελθόν πως ε, αν έχει κάποιος υπερβολικά μεγάλο ποσοστό της αγοράς ε, τελικά βλάβονται και οι καταναλωτές ε, γι' αυτό θα πρέπει να αποδίδουμε μεγάλη σημασία στον σωστό ανταγωνισμό. Και βεβαίω τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τις αρχές ανταγωνισμού που ανήκουν στο ευρωπαϊκό αυτοδίκτυο. Στόχος είναι όπως είπαμε, ο θέμητος ανταγωνισμός και η ορθότερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει με το να ακολουθούν κάποιες ελάχιστες κοινέ διατάξεις, ε, κάτι το οποίο θα οδηγήσει και σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ λοιπόν πως με βάση αυτά η πρόταση τη Κομισιόν επί τη αρχή πηγαίνει σωστή κατεύθυνση. Σε κάποια λίγα σημεία παρόλα αυτά θα έπρεπε να διορθωθεί. Το πρώτο είναι το σημείο 3 όπου αφορά το πώς θα εφαρμοστεί εδώ συγκεκριμένα η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συχνά το πρόβλημα ότι αυτό το οποίο αποφασίσαμε μετά δεν εφαρμόζεται σωστά. Και το ξανατονίζουμε και όταν διαπιστώνουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να ενισχυθούν ή να ξεκαθαρίσουν, θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο με μια παραπομπή στα εκτιμώντας, αλλά σεβόμενοι βεβαίως ε, τις αρμοδιότητες των κρατών μελών που είναι υπεύθυνα για την ε, διοίκηση, με κάθε σεβασμό, λοιπόν να προσπαθήσουμε να το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να είναι σαφές ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει συγκεκριμένη εφαρμογή και στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Γι' αυτό προτείνω να αναφερθούν ρητά τα α, οι σχετικές ε, διατάξεις ε, που αφορούν στο διοικητικό δίκαιο. Δηλαδή υπάρχει δικαίωμα να δει κανεί τον φακελό του, δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο, δικαίωμα να έχει μια δίκαιη δίκη, εμπιστευτικότητα με τον δικηγόρο του και βεβαίως ε, η δυνατότητα να γνωρίζει ποιο ακριβώς είναι αυτό το οποίο του καταλογίζει η εκάστοτε αρχή. Αυτά είναι αυτά τα οποία περιέχονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αφορούν ειδικά το δίκαιο του ανταγωνισμού. Το άλλο θέμα αφορά κάποια μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί και υπάρχουν στα εκτιμώντας ε, και εδώ πέρα τίνω να συμφωνήσω με την Κομισιόν, ε, δηλαδή το θέμα είναι το εάν εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα σήμερα ή όχι. Δεν σημαίνει λοιπόν πως αυτά τα πράγματα γίνονται αυτομάτως, γι' αυτό δεν υλοποίησα την αρχική μου σκέψη να βγουν αυτά κατευθείαν στο κείμενο, αλλά προσπάθησα τα μέτρα αυτά να είναι ένα στοιχείο των δυνατοτήτων της Κομισιόν. Ακόμα και αν είναι σαφές πως ε, η όροι βεβαίως που αφορούν τη μη επανορθώσιμη ζημιά είναι ένα πάρα πολύ υψηλό κατόφλι. Γι' αυτό θα ήθελα να γίνει μια μελέτη για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο και πώς μπορούμε να έχουμε ε, ενίως ευρωπαϊκούς κανόνες. Το τρίτο θέμα, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 11 ως υποχρεώσεις. Έχουμε λοιπόν υποχρεώσει αυτές οι οποίες αντικαθιστούν κάποιες απαγορεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού να έχουν επαρκείς πόρους για να μπορούν ακριβώ να εποπτεύουν τις υποχρεώσει και τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι διάφορες εταιρείε. Το τέταρτο σημείο, το οποίο είναι σημαντικό και είναι το πρώτο τελευταίο, αφορά το όριο των προστήμων του 10%. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε σωστούς όρους και ενιαίους όρους για τις επιχειρήσεις στην ενιαία ώρα. Οι αρχές συμφωνούν ότι ήδη το όριο αυτό είναι στο 10% άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην γίνει η ενιαία προδιαγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το πέμπτο και τελευταίο αγαπητοί συνάδελφοι είναι ακριβώς οι ε, αιτήσει αυτές οι οποίες, οι ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν ε, τους ε, βασικούς μάρτυρες και θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές εγγυήσεις και τα κίνητρα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να υπάρχει ταυτόχρονα βεβαίω, όπως είπα και η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ουσιαστικά σημεία της ε, έκθεσής μου. Να σας πω τώρα το χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, συζήτηση αυτών στις 20 Νοεμβρίου, έτσι ώστε μετά να ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου. Άρα λοιπόν ε, θέλω να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στους εισηγητές. Τι μπορούσαν για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πάντα θεωρούσαμε ότι είναι η Λιδία Λίθος μια ισχυρή πολιτική ανταγωνισμού, μια ε, ανταγωνιστική πολιτική για μια σωστή εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. Τον Ιανουάριο με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε μια έκθεση που είχα συντάξει εγώ ότι πρέπει να ενισχυθεί η αρχή ανταγωνισμού, να χρησιμοποιήσουμε όλε τι δυνατότητε που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή συνεργασίας. Σε επίπεδο S&D, στο μάσο σοσιαλιστών δηλαδή, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για αυτό το σχέδιο κειμένου και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αναφερθώ σε έξι σημεία. Δεν είναι εξαρτητικό ο κατάλογο βέβαια, αλλά είναι σημεία που θα επιβάλλουμε, επιβάλλουμε Θέλω όμω να αναφερθώ ε, σε αυτά. Δεν θα μακρηγορήσω. Πρώτα απ' όλα, όπως ήδη υπόθηκε στις ζητήσεις του Ιουλίου για μας, η ανεξαρτησία ε, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ανεξαρτησία ε, στην ηγεσία θέλετε, των εθνικών αρχών ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι πλήρης. Όχι μόνο απέναντι στις πολιτικές πιέσεις, αλλά θα πρέπει και η εκλογή τους ο ορισμός του να βασίζεται στην εμπειρία του, στα, πραγματικά του κριτήρια και όχι οποιαδήποτε άλλη πολιτική ε, διάσταση. Αυτό είναι που ε, καθιστά ανεξαρτήτη την αρχή. Επίσης δεν είναι συνεπής η έκθεση όταν μιλάει για προσβασιμότητα, accessible and in possession, προσβάσιμο και το in possession στο άρθρο 8 δεν είναι σωστό, διότι δίνει τη δυνατότητα σε κάποιε επιχειρήσει όταν δεν θέλουν να συνεργαστούν με τι αρχέ του ανταγωνισμού και δεν θέλουν να δώσουν πληροφορίε ε, να τι αποκρύψουν. Λέει, ότι δεν, δεν τα έχουν στην κατοχή δηλαδή δεν τα έχουν in possession. Επίση ε, πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση των αρχών ε, ανταγωνισμού δεν μπορεί να βασίζεται μόνο από τα πρόστιμα. Έχουμε κάποιε καλέ πρακτικέ σε κράτη-μέλη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ω παραδείγματα. Όμω θα πρέπει να είμαστε σαφεί εδώ. Τέταρτον, είμαστε πεπισμένοι ότι τα πρόστιμα αυτά πρέπει να βασίζονται στο παγκόσμιο τζίρο και όχι σε κάποιο άλλο σχετικό και ασαφές. Ε, επίσης, όταν μιλάμε για τους whistleblowers, εμείς πάντα υποστηρίζουμε τους whistleblowers πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μα να προστατεύσουμε. Μην ξεχνάμε όμω ότι ένα whistleblower δεν μπορεί ε, να είναι κάποιο ανταγωνιστή ή να έχει προσωπικό κέρδο, ε, διότι αυτό είναι αντιβαίνει τον αρχικό σκοπό του όλου εγχειρήματο. Πρέπει επίση να πω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει οι δημοσιογράφοι, πρέπει οι πολίτε να έχουν πρόσβαση στι πληροφορίες αυτές και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λαμβάνει και να μπορεί να συζητεί ε, τις αιτήσεις εκθέσεις όλων των ε, εθνικών ε, αρχών ανταγωνισμού. Να σας ευχαριστήσω καλή μια φορά Πρόεδρε ε, και τον εισηγητή για, την, για το σχέδιο έκθεσης. Θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, αυτό είναι βέβαιο, με τους, και με τους και εισηγητές και θα, θα διηγηθούμε ελπίζω στις κατάλληλες συμβαστικές λύσεις. Η τελική έκθεση θα είναι ακόμα καλύτερη και θα υπηρετεί ακόμα καλύτερα τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Από τη ΣΥΑΡ ο Ιν Σταμπάτη έχει το λόγο παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το ECR ε, βλέπει θετικά την πρόταση της Κομισιόν. Η πρόταση σέβεται τις διαφορές των κρατών μελών και αφήνει περιθώριο για τις εθνικές παραδόσεις Σέβεται δηλαδή την αρχή της επικουρικότητας. Αναλύσαμε την πρόταση του Ανδρέας Φαμπ και θα κάνουμε κάποιες προτάσεις. Το ECR έχει την εντύπωση πως η εναρμόνιση καυστομής δεν πηγαίνει αρκετά μακριά π.χ. Ε, θέλαμε να υπάρχει, ε, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, μια εναρμόνιση των εντολών, αλλά αυτό βεβαίως ε, μας βρίσκει κάπως αντίθετους, γιατί παραβιάζεται η αρχή της επικορικότητας. Κάποιες τροπολογίες επίσης αφήνουν κάποιο περιθώριο ερμηνείας, δηλαδή όταν τα πρόστιμα δεν αφορούν τον παγκόσμιο τζίρο αλλά τον σχετικό τζίρο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή όταν μιλάμε για τη σχετική αγορά, αυτό δεν έχει σχέση με το μέγεθος της επιχείρηση και την επιρροή που έχει στην αγορά. Έχουμε λοιπόν πολλά πράγματα τα οποία είναι στην διακριτική ευχέρεια και ήδη ακριβώ εδώ πέρα οδηγούμαστε στο να διαλέγει κανείς ρυθμιστικό καθεστώς, κάτι το οποίο υποτίθεται θέλουμε να εμποδίσουμε. Και λέει πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, το καθεστώς των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν τις ίδιες ε, δυνατότητες ε, με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται λογικό να λαμβάνεται υπόψη αυτό βεβαίως. Θα πρέπει να δούμε εάν η μεγάλη γκάμα προϊόντων αντικατοπτρίζει και ανάλογο μερίδιο της αγοράς και θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο. Συνολικά, το ECR ζητάει να ληφθούν υπόψη οι εθνικές διαφορές των κρατών μελών. Όλοι γνωρίζουμε ότι η υπερβολική εναρμόνιση σημαίνει μεγάλο κόστος προσαρμογής για τις εθνικές αρχές και τα πράγματα μετά αναβάλλονται ε, επάπειρον ε, ή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο λοιπόν καλά θα έκανε να προσανατολιστεί στο κείμενο που προτείνει η Κομισιόν. Και οι κύριε Σφάμπ οπωσδήποτε θα καταθέσουμε και τροπολογίες, αλλά συνολικά βλέπουμε με ενδιαφέρον και ικανοποίηση την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους τώρα ο Πίτερ Γιάτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Μάρκους. Η δική μου ομάδα υποστηρίζει ε, ιδιαίτερα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειαζόμαστε ελάχιστα κοινά πρότυπα για την έρευνα και, τις, ε, και τα εργαλεία κυρώσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, στο ΙΣΙΑ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει ένα πεδίο για τις εθνικές παραδόσεις θα μπορούσαν να συμφωνούσαν, μιλούσαμε για τον πολιτισμό. Αλλά εδώ όμως μιλάμε για ίσο ανταγωνισμό, για δίκαιο ανταγωνισμό, για εσωτερική αγορά και οι εθνικές παραδόσεις ε, δεν νομίζω να έχουν θέση εδώ. Εν πάση περιπτώσει, καλωσορίζω το γεγονό ότι ο εισηγητή θέλει να ενισχύσει κάποιε διατάξει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εποπτεία των αποφάσεων δεσμεύσεων ε, πρέπει να έχουν τα, τα απαραίτητα εργαλεία οι εθνικές αρχές για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με αυτές τις ε, απαιτήσει και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση να ξεκινάει μια διαδικασία παράβασης. Δεν είμαι τόσο βέβαιος βέβαια ότι κάποιες άλλες προτάσεις καθιστούν, βελτιώνουν το κείμενο της Κομισιόν ιδιαίτερα σε ό,τι φορά το αίτημα πληροφορίας σε ένα σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή θέλουμε οι εθνικές αρχές να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα ε, που να είναι προσβάσιμα και στις επιχειρήσεις. Όχι να είναι προσβάσιμα στις επιχειρήσεις, όχι να τα έχουν στη διάθεσή τους ίδιοι. Είναι κάπως ε, ξεπερασμένο να λέμε in their possession. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν την δικαιολογία ότι τις πληροφορίες δεν τις έχουν αυτοί, τις έχουν οι θηκατρικές τους κάπου αλλού, όταν γνωρίζουμε ότι η πληροφορία αυτή είναι απόλυτα προσβάσιμη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Επίσης ε, θα πρέπει οι αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στο cloud. Ακόμα και όταν μια τρίτη εταιρεία είναι αυτή που ε, για αυτά τα δεδομένα. Τώρα για τα πρόστιμα. Αντιλαμβάνομαι τον εισηγητή, ότι ο εισηγητής ε, λέει ότι πρέπει να είναι 10% το ανώτατο όριο σε σχέση με το τζίρο. Όμως αυτό δεν θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ε, τι εννοούμε όταν λέμε ε, το κατάλληλο, τζίρο, κατάλληλο relevant turnover, τι θα πει αυτό, είναι το ευρωπαϊκό τζίρο, ε, είναι ο τζίρος του καρτέλ. Ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως ε, που συχνά αποτελούν αντικείμενο ε, καταχρήσεων από τις μεγάλες επιχειρήσεις να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση θα πρέπει το πρόστιμο να αντικατοπτρίζει την πραγματική οικονομική ισχύ της επιχείρησης ε, η οποία ε, παραφέρεται. Δεν πρέπει να φορτωθούν σε μια θηγατρική εταιρεία και τα πρόστιμα στη συνέχεια να εξαφανιστούν. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντα θα έχουν πολύ χαμηλές πωλήσει σε σχέση με τις μεγαλύτερες ε, σε διεθνέ επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τι πληροφορίε που θα πρέπει να μοιράζονται οι εταιρείε με τους δικηγόρου τους και το δικαίωμα που έχουν οι εταιρείε ε, να μην ε, δέχονται ε, ότι έχουν ε, παραβεί τον νόμο όταν το, ζητάει η αρμόδια αρχή. Αντιλαμβάνομαι τι ανησυχίε του εισηγητή. Πρέπει να έχουν κάποια δικαιώματα επιχειρήσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτή η κατάλληλη προσέγγιση να το συμπεριλάβουμε. Δηλαδή, εδώ αυτό, αυτή την οδηγία. Αυτοί οι κανόνε εφαρμόζονται και ισχύουν ούτω ή άλλω σε όλου του τομεί του δικαίου. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε εδώ. Ε, χρειάζεται να διευκρινίσουμε περισσότερο από ό,τι αλλού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται δηλαδή και ειδική μεταχείριση εδώ στον τομέα του ανταγωνισμού. Το κεφάλαιο της αμοιβαία συνδρομής είναι ένα κεφάλαιο κλειδί. Χρειάζονται κοινέ εξουσίες οι εθνικέ αρχέ ακριβώς για να διευκολύνουν την ε, συνεργασία του Εγώ καλωσορίζω την πρόταση τη Κομισιόν στον τομέα αυτόν. βεβαίω αντιλαμβάνομαι κάποιε από τι αλλαγέ που θέλει να επιφέρει στο κεφάλαιο αυτό ο εισηγητή. Πρέπει όμω να εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα παρεμποδίσει τη συνεργασία μεταξύ των NCA, των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, την εκτέλεση των αποφάσεων, η εξαίρεση δεν πρέπει να επιτρέπει να μπορεί να επιληθεί με πρέπει να δώσουμε όλη τη δυνατότητα στην Κομισιόν να αξιολογήσει ε, το αίτημα από μια αρχή που, το, ε, που έχει αρνηθεί να ασχοληθεί με μια υπόθεση και να αφήσει αιτιολόγηση στην περίπτωση αυτή. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πέτερ από την ΚΟΕΙ Παλ, Παλώμα Λόπες Βερμέχο που δεν είναι εδώ. Ε, είναι εδώ η Μόλι όμως θα μιλήσει για τους πράσινους. Ε, ναι, πάλι θα... Τώρα θα είμαι ο Μισελ Ρόιμαν και μετά θα είμαι η Εύα Ζολή μετά από λίγο. Ε... Λοιπόν, για το σχέδιο έκθεση του κυρίου Σβάμπ, όπω και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη σημασία των προστήμων και το γεγονό ότι χρειαζόμαστε πρόστιμα στο κατάλληλο επίπεδο, έτσι ώστε να είναι πραγματικά αποτρεπτικά. Διότι αυτό είναι που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αποθαρρύνουμε τα καρτέλ. 10% λοιπόν του κατάλληλου τζίρου της επιχείρησης. Η πρόσθεση της Κομισιόν ήταν 10% του παγκόσμιου τζίρου. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό υπονομεύει την πρόσθεση της Κομισιόν, αυτό που προτείνει ο εισηγητής, διότι πρέπει να είναι αποτρεπτικά τα πρόστιμα και εμείς θέλουμε οι επιχειρήσεις να μην ξεκινήσουν καν αυτή τη διαδικασία να μπουν σε ένα κατέλ και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν όντως φοβούνται ότι το πρόστιμο θα είναι μεγάλο όταν τους πιάσουν. Ε, θα πρέπει λοιπόν το πρόστιμο να επί του συνόλου του τζίρου και να είναι τουλάχιστον 10%. Να υπάρχει δυνατότητα κράτη-μέλη να έχουν υψηλότερα ε, πρόστιμα εφόσον το επιθυμούν. Επίση, θεωρούμε ότι η αποζημίωση που θα πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση δεν, πρέπει, δεν θα πρέπει να ε, αφαιρείται από το πρόστιμο. Σε ό,τι αφορά τι δυνατότητε που θα έχουν οι αρμόδιε αρχέ να ζητήσουν στοιχεία. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο εισηγητή λέει ότι οι επιχειρήσει πρέπει να δίνουν πληροφορίε ε, προς τις εθνικές αρχές ε, εφόσον τις έχουν στη διάθεσή τους ενώ η Κομισιόν έλεγε πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μπορεί να φαίνεται μια λεπτή διαφορά αλλά είναι πιο περιοριστικό αυτό που προτείνει ο εισηγητής τα στοιχεία που βρίσκονται στο cloud ή που έχει μια άλλη που είναι στη διάθεσή της μια άλλη ε, θηγατρική είναι προσβάσιμα για την επιχείρηση αλλά δεν είναι στη διάθεσή της ε, δεν, θα πρέπει θα μπορούσε παραδείγματο χάρη κάποιο να δημιουργήσει μια θηγατρική για να ε, προχωρήσει σε ένα καρτέλ και όταν γίνει μια έρευνα αυτή η θηγατρική να μην έχει πληροφορίε στη διάθεσή τη. Και έτσι να μην χρειάζεται να τη μοιραστεί με τι αρχέ. Ε, κάποια άλλα σημεία όπου εμεί θα υποβάλουμε τροπολογίε, εμεί οι πράσινοι. Πρώτα απ' όλα θα προσθέσουμε ε, διατάξει για να αποφύγουμε σύγκρουση συμφερόντων στο άρθρο 4. Είτε με μια περίοδο μετάβαση όταν κάποιο φύγει από μία NCA ε, πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Όταν παραδείγματο χάρη υπάρχει κάποιο συγγενή ο οποίο ε, ε, εργάζεται σε μια εταιρεία που βρίσκεται υπό διερεύνηση. Ε, στο άρθρο 5 για του πόρου τώρα, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσουμε μια υποχρέωση για τα κράτη-μέλη ετησίω να αναφέρουν στην Κομισιόν του πόρου που έχουν στη διάθεσή του και η Κομισιόν να μπορεί να υποπτεύει του πόρου αυτού και αυτό θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε καθώς και δυνατότητα να επιβάλλει, να επιβάλλει συστάσεις. Επίσης θα προσθέσουμε μια διάταξη για την ανάγκη οι NCAs να αποφασίσουν αυτόνομα για τη χρήση του προπολογισμού τους. Τέλος, θέλουμε να διευκρινίσουμε το κεφάλαιο που αφορά ε, την leniency, δηλαδή την επίοικια. Ε, όταν αυτό αφορά τρεις χώρες και πάνω, η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για την υπόθεση αυτή και πρέπει να υπολογίσουμε και τον χρόνο για την ασυλία. Πρέπει να βασιστούμε εδώ στην πρόταση του συγκητή. Ευχαριστούμε τον συγκητή για το έργο του και ο Μισελ θα συνεργαστεί μαζί και τι τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ε, προτιμάμε την original ομιλήτρια, ό,τι ρόλο και αν παίζετε εσείς. Η Κάμπελ δεν είναι εδώ, η Γκίλ έχει ζητήσει το λόγο γιατί θέλει να φύγει. Νομίζω ότι δεν είχα χρόνο για catch Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή για την παρουσίασή του, για την έκθεσή του, συγγνώμη. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εθνικών αρχών για τον ανταγωνισμό και να ανοιχνεύονται οι παραβιάσεις του ανταγωνισμού. Είναι απαραίτητο να έχουμε όμως και τον κατάλληλο προϋπολογισμό για να το πετύχουμε αυτό. Πώς θα διασφαλίσουμε τους πόρους αυτούς και τα έσοδα που απαιτούνται. Και άλλοι συνάδελφοι έχουν θέσει το θέμα αυτό. Θα ήθελα να καταλάβω τη λογική σας σε σχέση με τα πρόστιμα. Πώς πιστεύετε ότι μια τέτοια μορφή επιβολής προστήμων θα λειτουργούσε στην αγορά με τη μορφή που έχει σήμερα. Είναι απαραίτητο να το γνωρίζουμε πριν εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει το λόγο. Λοιπόν, δίνω το λόγο για πολύ λίγο στον εισηγητή. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους συναδέλφους που μίλησαν ως σκιώδεις εισηγητές ή όπως είναι η Ναγκίλ ε, ως ανεξάρτητη συνάδελφος. Θεωρώ πως ε, πράγματι αξίζουν οι έπαινοι προς την Κομισιόν, αλλά πολλές από τις σκέψεις ε, που είδαμε να αναπτύσσονται ως κριτική με οδηγούν ακριβώς να σκεφτώ ότι η εκθεσή μου πηγαίνει σε καλή κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί επί της αρχής ότι θα πρέπει να ε, γίνουμε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για να δημιουργηθεί για όλους μια ασφάλεια δικαίου και ε, εντάξει, υπάρχει μια τάση εναρμονισμού, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαία αυτή η αγαπητέ συνάδελφε σε μια ενιαία αγορά. Για να υπάρχει και ίση μεταχείριση και των καταναλωτών. Το δεύτερο θέμα της ανεξαρτησίας της αρχής. Είναι και για μένα εξίσου σημαντικό όσο και για τους συναδέλφους, αλλά βεβαίως ε, είναι υπό τον ελέγχο των εθνικών κυβερνήσεων οι αρχές του ανταγωνισμού. Δεν αλλάζει αυτό δημοκρατικά. Έτσι είναι και πρέπει να ενισχυθούν οργανωτικά χωρίς βεβαίως να θίξουμε ακριβώς ε, την ιστορική οργάνωση των κρατών μελών. Οπωσδήποτε μπορούμε να αναζητήσουμε κάποιον συμβιβασμό στις διαπραγματεύσεις με τους συναδέλφους για το όριο των προστήμων ε, αναφέρθηκε πολλές ε, φορές ε, και χαίρομαι που οι συνάδελφοι προσανατολίζονται στο θέμα σχετική αγορά ή παγκόσμια αγορά και όχι στο 10% αυτό νομίζω το είχε ε, πει ο εκπρόσωπος των Πρασίνων Μόνο νομίζω όμως ότι εφόσον μιλάμε για μία ενιαία αγορά, λογικό είναι να μιλάμε γι' αυτό. Επίσης, στην συγκεκριμένη περίπτωση σχετική και παγκόσμια αγορά δεν θα πρέπει να σημαίνουν κάτι το διαφορετικό. Και τέλος, αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Γκίλ. Οπωσδήποτε θέλουμε οι πόροι των σχετικών αρχών να είναι επαρκής. Αλλά δεν μπορούμε να το καθορίσουμε αυτό ευρωπαϊκά. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος κάθε χώρας και την θέση βεβαίως της αρχής ε, στο πλαίσιο των θεσμών της ε, κάθε χώρας, αλλά είμαι διαθέσιμος να το συζητήσω για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία και τους πόρους των αρχών αυτών. Νομίζω και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την συνεισφορά τους. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Είπατε ήδη ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Μην τα ξαναλέω. Περνάμε στο σημείο 9 αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης. Ο Φούλβιο Μαρτουσέλο είναι ο εισηγητής. Έχετε τον λόγο, κύριε Πουλευτά. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή. Ελπίζω να παρουσιάζει ενδιαφέρον για όλους. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν ήδη 85 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να προσπαθήσω να ακούσω αυτά τα οποία λέγουν οι συνάδελφοι. Πολλές τροπολογίες συνεισφέρουν θετικά στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. γύρω από μια κατάσταση που χαρακτηριζόταν από μειωμένα επίπεδα αποτελεσματικότητας. Είναι σημαντικό να διευρυνθεί το πεδίο λοιπόν αυτό. Προβλέπονται να γίνουν σημαντικές τα έλεγα συζητήσεις γύρω από αυτό. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση έχει σχέση με τα ποσοστά τα οποία θα πρέπει να δοθούν στο κράτος το οποίο γίνεται η εκτέλεση. Εδώ η συζήτηση νομίζω ότι ήταν ήδη μέχρι τώρα πλούσια. Θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στο κράτος να διαχειριστεί πολλές φορές κάποιες διαδικασίες με υψηλό κόστος ε, το οποίο αυτό κόστος πρέπει να καλύπτεται βέβαια Υπάρχει το θέμα και της αξιολόγησης των ποινικών συνεπειών όπου γίνεται η κατάσχεση ή μάλλον η δίμευση των ποσών αυτών. Περιμένω προτάσεις ε, ενδιαφέρουσες στα πλαίσια της επόμενης συνάντησης των σκιωδών όπου θα προσπαθήσουμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Θα πρέπει να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση λοιπόν των ποινών και των διοικητικών αποφάσεων είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο αν θέλουμε οι εγκληματικές οργανώσεις να μην έχουν πλέον καύσιμο. Σας ευχαριστώ. Έρχομαι τώρα στους Κιώδης. Η Εύα θα αντικατοστήσει την Καταλίνα. Η Φόξ δεν είναι εδώ. Αλλά θα πάρει το λόγο Αφού διάβασα, λέει η κυρία Βίρινγκ, τις τροπολογίες σας και την πρότασή σας, να υπογραμμίσω ότι έχει μεγάλη σημασία η απόφαση αυτή για την ασφάλεια μακροπρόθεσμα των πολιτών μας. Πρέπει όμως να ε, διασώζουμε και τα δικαιώματά τους. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια βιώσιμη λύση εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες ασφαλείας. Το μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους συναδέλφους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ είναι σαφές. Πιστεύουμε ότι ο κανονισμός αυτός πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα νομικά μέσα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τις αρχές της ε, δικαιοσύνης και για τα μέλη και για τα κράτη-μέλη. Ε, το κράτος μέλος το οποίο εκδίδει την απόφαση πρέπει να παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι της ποινή που επευλήθηκε για λόγους εγκληματικών ενεργειών αλλά θα πρέπει να καλύπτεται και το κόστος για τα κράτη τα οποία εκτελούν την κατάσχεση. Συνεπώς λοιπόν η καλύτερη λύση είναι να δίδουμε στην χώρα που εκτελεί την απόφαση ένα τμήμα της ποινή του κέρδους αν θέλετε, για να καλύψει το κόστος. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι σε σχέση και με τις χρονικές προθεσμίες Δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε την πρόταση, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και πρέπει να παραμείνουμε φιλόδοξοι κατά τη διάρκεια της πρότασης. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο αποστέλουμε προς το Συμβούλιο. Γιατί όλοι τελικά τον ίδιο στόχο έχουμε, να μην χρηματοδοτούνται οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην πηγή, να έχουμε τους απαιτούμενους πόρους και τότε θα πετύχουμε. Ευχαριστώ. Η Εύα θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ εκ μέρους του συναδέλφου του κύριου Κάτλιν να πω ότι εμείς συγχαίρουμε τον εισηγητή για το έργο του. Πρέπει να υπάρξει μια επιτάχυνση να σημειωθεί γρήγορη πρόοδος ε, σε ό,τι αφορά την ανάκτηση ε, προϊόντων εγκλήματος σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Ε, θα πρέπει βεβαίως να φέρουμε στη δικαιοσύνη τους ενόχους υπεύθυνους, αλλά το βασικό είναι η ανάκτηση των προϊόντων εγκλήματος. Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των δικαστηρίων, είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να να περιβάλλεται από εμπιστοσύνη το σύστημα το ευρωπαϊκό. Είναι πάνω από 120.000 ευρώ το όριο ε, σε ό,τι αφορά Όταν είναι πάνω από 120.000 μάλλον ευρώ το, το ποσό ε, για την εκτέλεση θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει μεταβίβαση. Στο άρθρο 3 είναι ε, ο κατάλογος εξαντλητικός, η Κομισιόν μέσα από πλάξη επικαιροποιημένα τακτικά, θα έχει τον κατάλογο των αδικημάτων που θα καλύπτονται και βεβαίως αναμένουμε ανεπομονησία τη συζήτηση για τις τροπολογίες στην επόμενη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Μόλι θα γίνει Εύα. Ε, ε, ναι, την Εύα Ζολή εγώ βέβαια εκπροσωπώ, να μην μπερδευτούμε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, για τον, τον εισηγητή μάλλον για το κείμενο, έχουν γίνει μια σειρά προτάσει βελτίωση και θέλω να πάμε κάπως πιο μακριά σε κάποια σημεία. Επίσης είμαστε υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου. Η Κομισιόν προ... αναφέρει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων για τις ποινικέ διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχει όμως αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων που παίρνονται και στα πλαίσια διοικητικών ε, διαδικασιών όταν αυτές συνδέονται με ποινικέ υποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών. Ε, όταν ένα ποινικό δικαστήριο παίρνει την απόφαση δέσμευση ή δίμευση, εμεί είμαστε υπέρ και των διοικητικών ε, προληπτικών διαταγών, όπου η δίμευση μπορεί να γίνει όταν δεν μπορεί κάποιο να αποδείξει την προέλευση κάποιων προϊόντων. Εφόσον βεβαίω γίνονται σεβαστά τα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε επιβάλει τροπολογίε για να διευρυνθεί επίση το πεδίο των αδικημάτων να καλύπτονται και τα προϊόντα από φοροποφυγή και φοροδιαφυγή. Ε, στο άρθρο 3 έχουμε ένα κατάλογο, συμφωνούμε με τις λοιπές οικονομικές, ε, τα οικονομικά αδικήματα που προλαμβάνει ο εισηγητής, θέλουμε να προσθέσουμε όμως και τα φορολογικά αδικήματα, φορολογική απάτη ε, και φοροποφυγή, φοροδιαφυγή. Βεβαίως κάποιες χώρες ε, δεν στέλνουν τρία χρόνια στη φυλακή ε, τα, τους παραβάτες για τέτοιες, ε, τέτοια αδικήματα, ίσως θα πρέπει να το ευθυγραμμίσουμε στα δύο χρόνια, γιατί αυτό ισχύει στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα, την ανάκτηση των προϊόντων εγκλήματος, όταν έχουμε πάνω από 10.000 ευρώ, το κράτος το οποίο έχει εκδώσει την διαταγή και αυτό που το εκτελεί θα πρέπει να μοιραστούν το ποσό. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι διαφορετική η προσέγγιση. Όταν το ποσό είναι πάνω από 10.000 ευρώ τα 10.000 θα πρέπει να δίδονται στη χώρα εκτέλεση για να καλυφθεί το κόστος εκτέλεση τη δίμευση και το υπόλοιπο ποσό πρέπει να πανέχεται στη χώρα που έχει εκδώσει τη διαταγή. Αυτό προτείνουμε εμεί, Ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία τώρα. Θα προτείναμε τα κράτη-μέλη να μοιράσουν τα στατιστικά στοιχεία για τι διαταγές δίμευση κάθε 6 μήνες και όχι κάθε χρόνο με την Κομισιόν, έτσι ώστε η Κομισιόν κάθε χρόνο να εκδίδει μια έκθεση που αναλύει τα στατιστικά στοιχεία αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση, θα προτείναμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί τον κανονισμό αυτό σε 3 χρόνια από τώρα αντί για 5 χρόνια. Αυτά. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή και βεβαίως αναμένουμε μια... και προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω κάποιον άλλον, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να ζητήσει τον λόγο. Λοιπόν, Φλάβιο, Φούλβιο, θέλετε να προσθέσετε κάτι, να συνοψίσετε αυτό τα οποία είπαν συνάδελφοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπαμε είναι πλούσια και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εδώ καταγράφονται θα έλεγα συμφέροντα τα οποία ρυθμίζονται από τα συντάγματα των κρατών χωρών. Νομίζω ότι στα πλαίσια των συζητήσεων του σκιωδών θα καταλήξουμε, θα γεννήσουμε λέει ο μιλητής ένα ενδιαφέρον κείμενο Ελπίζω οι τροπολογίες να είναι ενδιαφέρουσες και στην Ολομέλεια να φτάσει ένα κείμενο το οποίο θα ψηφιστεί από την πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αν έρθετε αύριο το πρωί θα έχει αλλάξει η διαρρύθμιση γιατί θα έχουμε τις ακροάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια το απόγευμα. Οπότε θα είναι αλλού η θέση σας, αλλά έχετε θέση να ανησυχείτε για την έκθεση αυτή, το ξέχασα, ψηφοφορία στην Επιτροπή 6 Νοεμβρίου και θα δούμε μετά εάν Α, η Λίμπε θα ψηφίσει Δεκέμβριο-Ιανουάριο και θα δούμε μετά πότε θα πάει στην Ολομέλεια. Λοιπόν, αύριο άρα καθόμαστε διαφορετικά. Λίγα τη συνεδρία, ευχαριστώ.